La séance est ouverte. Συνάδελφοι, ξεκινάμε. Οπότε παρακαλώ να σταματήσουν ε, οι κατηδίαν συζητησούλε. τα πηγαδάκια. Παρακαλώ πολύ. Σα θυμίζω ότι ξεκινάμε με τις ψήφους. Ξεκινάμε τις ψηφοφορίες. Είναι περίπλοκη η διαδικασία. Έχουμε προετοιμάσει την πολιτική διάσταση αυτών των ψηφοφοριών στην συνάντηση των συντονιστών χθες το βράδυ. Οπότε ε, είμαστε κατά βάση σίγουροι ότι ε, τα, οι ψηφοφορίε θα γίνουν με πλήρη διαφάνεια. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Βέβαια, από τεχνική πλευρά πάντω έχουν ρυθμιστεί τα πράγματα. Πρώτον, Ε, κοιτάξτε να είστε σίγουροι ότι έχετε την κάρτα σας, την ηλεκτρονική σας κάρτα για την περίπτωση που θα χρειαστεί να ψηφίσουμε ε, ονομαστικά. Δεύτερον, θα ήθελα να ζητήσω από το συντονιστή του ΕΛΚ ε, να μου, να μου πει αν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, αν έχουμε δηλαδή απαρτία ή όχι. Ο Σαλβαντόρ δεν έχει την κάρτα του, ε. Υπάρχουν συνάδελφοι που έφυγαν να πάνε να ψάξουν την κάρτα τους. Οκ, θα τους περιμένουμε λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι όλοι μπορούν να ψηφίσουν. Μετά. Έχετε μπροστά σας παρακαλώ ε, τις, τους καταλόγους ψηφοφοριών. Ο τελευταίος ε, ετοιμάστηκε, τυπώθηκε πριν από μερικά λεπτά. Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση της Φραντσέσκα Μπαρτσάνη. Είναι η εντολή για τον τριμερή διάλογο. Tout le monde est au point. Όλοι έτοιμοι. Θα ξεκινήσουμε να ψηφίσουμε διανατάσεις τη της ε, χειρός και κάποια στιγμή θα χρειαστούν και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες βέβαια. Διανεμήθηκαν οι κατάλογοι ψηφοφοριών. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Ξεκινάμε, θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες διανατάσεως χειρός και μετά από μερικά λεπτά όταν όλοι έχουμε στα χέρια μας τις ηλεκτρονικές μας κάρτες, αν χρειαστεί, θα κάνουμε και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Η συγγήτρια είναι έτοιμη. Όχι. Bien. Alors, le rapporteur... Λοιπόν, συγγήτρια έτοιμη, όλοι έτοιμοι. Οπότε, ξεκινάμε να ψηφίσουμε τις τροπολογίες για την έκθεση Μπαλτσάνη. Πρώτη τροπολογία, ε, συμβαστική τροπολογία α, υπέρ. Κατά. Μία ψήφος κατά αποχές. Καμία αποχή. Γίνεται δεκτή η πρώτη συμβαστική πρόταση. Περνάμε στη συμβαστική πρόταση Β της συγγήτριας. Ε, έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία από τους φιλελεύθερους. Ο συμβασμός χωρίς τη φράση και πιστεύει ακράδαντα ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να τη χάνουν εγγύσεων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Ποιος είναι υπέρ αυτού του πρώτου τμήματος. Ευχαριστώ. Κατά. Μία ψήφος. Δύο ψήφοι. Τρεις ψήφοι. Τέσσερις κατά. Α, αποχή ήταν οι δική σας. Οκ. Okay. Δύο κατά και δύο αποχές. Μετά, δεύτερο τμήμα που προσθέτει αυτό το κομμάτι της φράσης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Η φιλελεύθερη, η συντηρητική και η κυρία Ανδρέασεν. Είναι όμως μειοψηφία. Οπότε και το δεύτερο τμήμα υιοθετείται. Περνάμε στην τροπολογία Γ. Υπέρ. Συμβαστική τροπολογία Γ. Υπέρ. Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Υιοθετείται. Συμβαστική πρόταση D. Υπέρ. Κατά. Τέσσερις. Πέντε. Πέντε ψήφοι κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Υιοθετείτε. Τροπολογία, συμβασική τροπολογία Ι, ε, υπέρ. Κατά. Τέσσερις ψήφοι κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Συμβαστική τροπολογία F. Υπέρ. Κατά. Καμία ψήφος κατά. Αποχές. Μία αποχή. Υιοθετείτε. Συμβαστική τροπολογία G. Υπέρ. Κατά. καμία αποχές, μία αποχή. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία H. Υπέρ. Κατά. Ναι, λίγο περισσότερο αυτή τη φορά. Αποχές. Καμία αποχή. Έξι ψήφι κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία I, J, υπέρ. Οι τι κάνουν, υπέρ. Κατά. Δύο ψήφοι κατά, αποχές. Καμία αποχή εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία J, υπέρ κατά τρεις ψήφοι κατά αποχές καμία αποχή εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία K κάπα υπέρ υπέρ είπα κατά πρέπει να μετρήσουμε νομίζω οι, αυτοί που είναι κατά παρακαλώ να κρατήσουν το χέρι τους ψηλά. Αποχές. 9 ψήφοι κατά αποχές. Υπέρ. Υπέρ τελικά το αποτέλεσμα. Διοθετείτε. Μετά περνάμε στις υπόλοιπες τροπολογίες. Τροπολογία 7. James Ellis. Η εισηγήτρια είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Όλοι οι υπόλοιποι. Αποχές. Τρεις αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Και πάλι James Ellis. Η συγκίτρια είναι κατά. Υπέρ. Τέσσερις ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Μιγγέλ Πόρτας. Ε, για διαγραφή. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιος ψηφίζει υπέρ. και πόρτας βέβαια, κατά, πολύ, αποχές, καμία αποχή, απορρίπτεται. Τροπολογία παριθμών 10 της κυρίας Ανδρέας, η συγγήτρα είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Καμία αποχή. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Λαβία. Που συμπεριλαμβάνει μια προφορική τροπολογία. Για να προσθεθεί economic and social. Οικονομικό και οικονομικό πριν αύξηση. Ο συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Κανείς. Αποχές. Ομόφωνα εγκρίνεται. συγχαίρουμε την ε, υποβάλλουσα την τροπολογία. 12. Τροπολογία 12. Α, έχει καταπέσει. Γιατί οθετήθηκε συμβαστική πρόταση Α. Το ίδιο και η 13. Φτάνουμε στην 20. Όλες οι άλλες έχουν καταπέσει. Από τη 12 μέχρι τη 19. Τροπολογία 20 του κυρίου Κλούτε. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιος ψηφίζει υπέρ. Είπα η συγκεκριμένη συμφωνεί. Κατά. Ηλεκτρονική ψήφος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχω δικαίωμα να ψηφίσω. Άρχεται η ψηφοφορία. Προσπαθούμε να την ξεκινήσουμε. Κλείνει η ψηφοφορία. 13 ψήφοι υπέρ, 19 κατά. Υπάρχει μία ψήφος ακόμα που δεν είναι ηλεκτρονική, μία ψήφος κατά που δεν είναι ηλεκτρονική, έτσι και, και μία ψήφος υπέρ που δεν είναι ηλεκτρονική, οπότε απορρίπτεται. Περνάμε στην 21, καλύπτεται από την ε, συμβαστική πρόταση Β. 22, ο Τζοβάνι Λαβία, ποιος είναι υπέρ, η συγγήτρια συμφωνεί. Κατά. Δύο ψήφοι κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23. Με δύο συγγραφείς. Με προφορική τροπολογία Α, μάλιστα. Υπάρχει την προφορική τροπολογία της ηγετρίας που προτείνει να μεταφέρουμε αν, την τροπολογία αυτή αν υιοθετηθεί στην παράγραφο 23α. Τώρα, επί της ουσίας, που προέρχεται από την Επιτροπή ΙΜΚΟ, η ηγέτρια είναι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Μ, αρκετή. Πέντε. Αποχές. Μία αποχή. Λοιπόν, η, η πλειοψηφία είναι υπέρ, υιοθετείται η τροπολογία και η, η συγγήτρια προτείνει να ενταχθεί στην παράγραφο 23α. Προφορική τροπολογία της Φραντσέσκα Μπαλτσάνη να αντικαταστήσει το συν 3,6% με το συν 4,7% στην παράγραφο 4 μια μικρή λεπτομέρεια που αντιπροσωπεύει μερικές εκατοντάς εκατομμύρια. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Πέντε. Αποχές. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Ε, οι τροπολογίες υποσημειώσεις ε, καταπίπτουν μάλλον στο κάτω μέρο της σελίδα καταπίπτουν, οι τροπολογία στο πάνω μέρος τη επόμενης σελίδα. Επίσης φτάνουμε στην 29 Χάρτονγκ. Ποιο είναι υπέρ, η συγγήτρια διαφωνεί. Δύο είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. αποχέ. Απορρίπτεται. Στο τροπολογία 30, James Ellis, η συγγήτρια συμφωνεί. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Κανεί απόχέ. Συγχαρητήρια στον James Ellis. Η τροπολογία του υιοθετήθηκε. Ε, οι επόμενες ε, μέχρι την 45 καλύπτονται. Φτάνουμε λοιπόν 45 James Ellis. Εδώ διαφωνεί η συγγήτρια. Ποιος ψηφίζει υπέρ. Τρεις. Κατά. Ωραία, πλειοψηφία, αποχές, κανείς, απορρίπτεται. Τροπολογία 46 των φιλελεύθερων. Η συγγήτρια συμφωνεί. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Μία ψήφος μόνο. Αποχές. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. 47 των ίδιων. Ε, και η συγγήτρια συμφωνεί και εδώ. Υπέρ. Κατά. Τέσσερις ψήφοι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη 48 και τη 49. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μία-μία. 48 του κυρίου Άρτονγκ. Διαφωνεί η συγγήτρια. Ποιο είναι υπέρ. Κύριε Αντρέασεν. Και ο κύριο Μοργκάντη. Δύο. Κατά. Πλειοψηφία. Αποχές. Καμία αποχή. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 49 των κυρίων Άγγλων και Φερχόφστατ. Η συγγέντρια συμφωνεί. Ποιο ψηφίζει υπέρ. Κατά. Μία ψήφο. κατά. αποχέ. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Υιοθετείται. Περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 50. Πληροφορούμε ότι αυτή η τροπολογία θα έπρεπε να αφορά... Ναι, λοιπόν υπάρχει μια γραπτή τροπολογία 50 και μια προφορική τροπολογία του Τζοβάν Λαβία. Και όπως και σε μια προηγούμενη προφορική τροπολογία, αν υιοθετηθεί ή 50, άνιοθετηθεί. αν υιοθετηθεί η προφορική τροπολογία θα ενταχθεί στην παράγραφο 13. Οπότε, ψηφίζουμε την 50 με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές, 8 ψήφι κατά, μία αποχή. Πλειοψηφία υπέρ. Τροπολογία εγκρίνεται και θα τοποθετήσει στην παράγραφο 13. Οι επόμενες τρεις τροπολογίες καταπίπτουν. Φτάνουμε στην 54. James Ellis, η εισηγήτρια διαφωνεί. Ποιος ψηφίζει υπέρ. Έντεκα. Κατά. 17. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 55. Γκέραν Φέρμ. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος ψηφίζει υπέρ. Κατά. Μία ψήφο. Δύο ψήφοι κατά. Α, τρεις. Αποχές. Καμία αποχή. Υιοθετείται. Τροπολογία 56 της Μάρτα Αντρέασεν. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιος ψηφίζει υπέρ. Η κυρία Αντρέασεν, κατά. Αποχές. Μία αποχή. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57 των κυρίων Χάγκλον και Φερχόφστατ. Η συγγήτρια διαφωνεί. Ποιος υπερψηφίζει. Η φιλελεύθερη και η κυρία Αντρέσεν. Κατά. Μια πλειοψηφία, αποχές, Δύο εποχές απορρίπτεται. Τροπολογία Χάρτονγκ 58. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιος φύζει υπέρ. Μία ψήφος υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 59. Λάγιος Μπόκρος. Που συμπίπτει με την 60 της κ. Τρούπελ και την 61 του κυρίου Μοργκάντη. Η συγγήτρια διαφωνεί. Ποιος είναι υπέρ αυτών των τροπολογιών. Που είναι ταυτόσιμες. 11. Κατά. Σηκώστε το χέρι σας παρακαλώ. 16. Αποχές. Απορρίπτονται αυτές οι τρεις τροπολογίες. Τροπολογία 62 των κυρίων Χάγκλουντ και Φερχόπστατ. Και εδώ η συγγήτρια προτείνει, αν υιοθετηθεί η τροπολογία, να ενταχθεί σε μια καινούρια παράγραφο 14α. Επίσης, η συγγήτρια έχει ζητήσει ψηφοφορία, χωριστή ψηφοφορία σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα που ξεκινάει από το observes, παρατηρεί και τελειώνει στο of budget 2000, ε, του προεπισμού 2011. Η γιατί διαφωνεί. Ποιος είναι υπέρ. Επτά. Κατά. Πλειοψηφία. Αποχές. Μία αποχή. Το πρώτο τμήμα καταπίπτει λοιπόν. Δεύτερο τμήμα. In this context, έτσι ξεκινάει, μέχρι το clear difference to the EU annual budget. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονική ψήφος. Θα συμμετάσχω εγώ στην πληροφορία, μπορώ. Αν το επιτρέπει η ομάδα μου. Ε, άρχεια ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. 17 ψήφοι υπέρ, 16 κατά. 18 υπέρ. 18 υπέρ. 16 κατά. Σαλβαδόρ, έχει την κάρτα σου πια, άρα μετρήθηκε. Ε, άρα υιοθετείτε αυτό το δεύτερο τμήμα. Τρίτο τμήμα. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιο ψηφίζει υπέρ. Πέντε. Κατά. Πλειοψηφία. Αποχές. Το τρίτο τμήμα απορρίπτεται. Οπότε, από αυτή την 62 κρατάμε το δεύτερο τμήμα το οποίο θα ενταχθεί σε μια καινούρια παράγραφο την 14α. Έτσι κύριε Συγήτρια, πολύ ωραία. 63. James Ellis. Η συγγήτρια διαφωνεί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Πλειοψηφία. Αποχές. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται. 64. Λούκα Άρτογκ. Η συγκίτρια διαφωνεί. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχέ Απορρίπτεται. Τροπολογία 65 του κυρίου Χάγκλοντ. Η συμφωνή. συμφωνεί. Ποιος άλλος είναι υπέρ. Κατά. Κανεί αποχές. Συγχαρητήρια τον κύριο Χάγκλοντ. Ομοφωνία υπέρ. Τροπολογία 66. Μοργάντη αφορά μια διαγραφή. Η συγκήτρια διαφωνεί Ποιο είναι υπέρ. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 67. Κύρια Ματέρα. Α, ε, έχει αποσυρθεί, δεν θα την ψηφίσουμε. 68. Μπόκρο. Η συγκήτρια είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. 3. Κατά. εποχέ. απορρίπτεται. 109 Χαρτόγκ, κατά ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία ε, του κυρίου Μπόκο, ποιο είναι υπέρ. Κατά και την 70. Τρόπο, ε, αποχές Δύο εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 71. Τζοβάνι Λαβία. Η συγητής υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υπέρ είναι η πλειοψηφία. Εγκρίνεται. 72. Έλγα Τρούπελ. Η συγητής υπέρ. Υπέρ. Αποχέ. αποχές απορρίπτεται 73 καλύπτεται 74 Κλάδιο Μοργάντη εισηγητής κατά ποιος είναι υπέρ 2 κατά μεγαπλειοψήφια αποχές απορρίπτεται 75 Δελαβία υπέρ κατά 7, 8, αποχές, εγκρίνεται. 76 Triple Τρίπελ. Εισηγητής είναι κατά πίσουν υπέρ. Κατά. Αποχές μία αποχή, απορρίπτωτα. 77, ε, Helga Trippel. Η συγγετής είναι κατά, υπέρ, 3, κατά. Η πλειοψηφία αποχές Απορρίπτωτα. 78, Μπόκρος. Η συγγετής είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. 4, κατά. Οι περισσότεροι αποχές 2. Απορρίπταται. 79 Χάγκλουντ. Εισηγητή κατά. ποιο είναι υπέρ. Πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχο Για την 79 του κυρίου Χάγκλουντ. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. 20 υπέρ, 16 κατά μία αποχή. Δύο αποχές. Λοιπόν, εγκρίνεται 80 τρίπελ. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Θα υποχρεωθούμε να κάνουμε και εδώ ηλεκτρονικό έλεγχο, γιατί μεγάλες ομάδες ε, έχουν διαρρεθεί. 80 τρίπελ. Ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικό έλεγχο. Τέλο. Αποτέλεσμα 21 ψήφι υπέρ, 22, 16 ψήφοι κατά. Η Έλγα Τρίπελ λοιπόν ε, περνάει την τροπολογία τη. Είναι συμβατή με το 81 του κυρίου Χάγκλοντ για την ίδια παράγραφο. Οπότε ψηφίζουμε την 81 με την υποστήριξη του εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Πέντε. Αποχές. Μία. Άρα εγκρίνεται η 81. 82. Ο εισηγητής προτείνει να εγκριθεί να γίνει μια νέα παράγραφος 76α. Ο εισηγητής είναι υπέρ αυτής της 82. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Τρεις. Αποχές. Μία. Εγκρίνεται. Θα μπει μία παράγραφος 76α νέα. Τροπολογία 83. Χάρτογκ. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ? Ένας. Δύο ψήφοι υπέρ. Κατά αποχές δεν υπάρχουν, απορρίπτεται 84 Χάγκλουντ με προφορική τροπολογία διαγράφεται η λέξη that είναι υπέρ οι εισηγητής ποιος είναι υπέρ κατά αποχές μία αποχή και μία ψήφος κατά εγκρίνεται με την προφορική τροπολογία 85 κλούτε κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Με την προσθήκη της λέξης Δίπλη. Ο εισηγητής είναι κατά πίσω υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η λέξη deeply. Δεύτερο τμήμα με την προσθήκη της λέξης social. Υπέρ υπέρ της λέξης social. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη λέξη social. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Αποτέλεσμα. Υπέρ της λέξης κοινωνικός 15, 16 ψήφοι, κατά 22. Η λέξη social λοιπόν διαγράφεται. βλέπει ο κόσμος ότι η Επιτροπή Προπολογισμών καταστρέφει το κοινωνικό το σώσα. Λοιπόν, τροπολογία 86. Μπάρμπαρα Ματέρα. Δύο τμήματα και εδώ. Πρώτο τμήμα. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Οκτώ αποχές. Η πλειοψηφία είναι υπέρ. Δεύτερο τμήμα. Εξηγητή είναι υπέρ. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα και γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Γίνεται 86. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. 14 ψήφοι υπέρ. 23 ψήφοι κατά συν μία ψήφο. οπότε απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Πάμε μετά στην τροπολογία 90, οι άλλε καλύπτονται, πόρτας, η συγγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ? Η Γκουέ. Κατά. Άποχες. Η πλειοψηφία είναι για την απόρριψη. 91. Από την Επιτροπή Μεταφορών. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας Επιτροπής Μεταφορών κατά. Δύο ψήφοι κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92 Χαρτόγκ. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Μία ψήφο υπέρ. Κατά. Οι υπόλοιποι αποχές απορρίπτεται. 93 Μοργάντι. Η συγγήτρια είναι κατά. Υπέρ. 4-5 κατά οι περισσότερες αποχές απορρίπτεται τροπολογία 94 με πολλούς που την έχουν υπογράψει από πολλές ομάδες και πολλές εθνικότητες η συγγήτρια είναι υπέρ υπέρ κατά τέσσερις αποχές εγκρίνεται 95 Χάγκλουντ αποσύρεται 96 η συγγήτρια είναι κατά υπέρ μας διαιρεί αυτή η τροπολογία οπότε η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 96 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. «22 ψήφοι υπέρ, συν μία ψήφος 23, 14 ψήφοι κατά και εγκρίνεται η τροπολογία». Πάμε στην 97 του κυρίου Μπόκρος, που είναι ταυτόσημη, με την 98 του κυρίου Χάρτονγκ. Η εισηγήτρια είναι κατά. Υπέρ. 4. Κατά. Οι περισσότεροι αποχές απορρίπτονται οι δύο 99 της κυρίας Ανδρέασαν. Η συγγήτρια είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Απορρίπτεται. Τροπολογία 100 της Επιτροπής Μεταφορών. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά μία ψήφος. Κατά αποχές, δύο αποχές, τρεις αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 101, διαφόρων συντακτών, η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Δύο αποχές δεν υπάρχουν, εγκρίνεται. 102 της Επιτροπής Μεταφορών, αλλά εδώ η συγγήτρια δεν τη θέλει. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία. Αποχές. Τρεις αποχές. Τέσσερις αποχές. Πέντε αποχές. Απορρίπτεται. 103. Μπόκρος. Η συγκήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Τρεις κατά οι περισσότεροι αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 104 Χάγκλουντ. Η συγκίτρια να καταπίσουν υπέρ. 4 κατά αποχές απορρίπτεται. 105 Ματέρα. Η συγκίτρια είναι κατά. πίσω υπέρ. Κατά. Άποχες ομοφωνία κατά της Μπάρμπαρα. Εκπληκτικές σκηνές αυτές. Λοιπόν, απορρίπτεται η τροπολογία. 106 του κυρίου Χαρτόγκ. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ? Ένα. Κατά. Η πλειοψηφία αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 107 του κυρίου Λαβία. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά να κρατάτε τα χέρια ψηλά όσοι είσαστε κατά. Κατά λέμε. Οκτώ. Εννέα κατά αποχές. Η πλειοψηφία είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 108 του κυρίου Χάρτονγκ. Η συγκήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Ένας. Κατά. Η πλειοψηφία αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 109 Helga Triple. Η συγγήτρια είναι κατά. Υπέρ. Δέκα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110 Καλ Χάγκλουντ. Η συγγήτρια είναι κατά. Υπέρ. ίδιο σχετισμό ψήφων σχεδόν, κατά. Θέλετε να κάνουμε επαλήθευση. Όχι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Αποχές απορρίπτεται και αυτοί. 111 Λούκας Χάρτογκ. Η συγκήτρια είναι κατά υπέρ. Κατά. Μεγάλη πλειοψηφία. Αποχές απορρίπτεται. 112 Χέλκα Τρίπελ. Η συγκήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. 6. Κατά αποχές απορρίπτεται. 113 μπόκρος υπέρ. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. 7 κατά. Η πλειοψηφία αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 114 του κυρίου Χάγκλουντ. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Έντεκα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 115 Τζοβάνι Λαβία. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. αποχές ήδη σχετισμός ψηφών όσον αφορά την παράγραφο 31 αλλά αυτή τη φορά η τροπολογία 115 γκρίνεται. 116 Μοργάντη η είναι κατά ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτωτα 117 Συντόνια και κάποιοι συνάδελφοί τη Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. άποχε. Εγκρίνεται. 118. Μάνερ Χάγκλουντ. η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Μία ψήφο, Κατά άποχε, εγκρίνεται. Είναι συμβατή με την 119 του Μιγκέλ Πόρτα. Η συγκίτρια είναι επίση υπέρ. Υπέρ της 119 ποιος είναι. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120 του κυρίου Χάγκλοντ. Η συγγήτρια είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 121. Χέλγα Τρίπελ. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Η πλειοψηφία αποχές απορρίπτεται. 122 του κυρίου Μοργάντη. Η είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 123 του κυρίου Λαβία. Στην αρχική παράγραφο έχουμε προφορική τροπολογία να αντικατασταθεί το reshuffle με το simplify. Και παροτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τον προβληματισμό της σχετικά πώς να απλουστεύσει το περίπλοκο σύστημα simplify και όχι reshuffle. Διευκρίνηση σημαντική. Εισηγείται εν υπέρ της τροπολογίας και της προφορικής τροπολογίας. Ποιος είναι υπέρ, κατά, δύο Δεν θέλετε να απλουστεύσετε εσεί οι συντηρητικοί, ε. Αποχές. Και οι πράσινοι δεν θέλουν τίποτα. Ούτε μεταρρύθμιση, ούτε απλούστευση. Πλειοψηφία υπέρ της 123. 124 Μόνικα Χολμάιερ. Εισηγήτριαν υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Κανείς, αποχές, η Μόνικα ομόφωνα. Οπότε της φυλά το χέρι ο πρόεδρος. Τροπολογία 125. Καρλ Χάγκλοντ. συγγήτρια κατά. Ποιος είναι υπέρ. Επτά. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 126 της κυρίας Γέγκλε. Η είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Τρεις. κατά. Τέσσερις μάλλον. Οι περισσότεροι είναι κατά. Απορρίπτεται. 127 μπόκρος. Η είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Τέσσερις. κατά. Οι περισσότεροι απορρίπτεται. 128 γέγκλε. Η συγγήτρια είναι υπέρ αυτή τη φορά της 128. Ποιος είναι υπέρ της 128. Κατά. Τρεις. Αποχές. Δύο. Εγκρίνεται 128. 129 Helga Triple. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να γίνει ηλεκτρονικό έλεγχος για την 129. Συγγήτρια είναι υπέρ. Ψηφίζουμε την 129 ηλεκτρονική ψηφοφορία που ξεκινά τώρα. Ψηφίσατε όλοι. τέλο 15 σε μία ψήφος 16, 23 ψήφοι. Κατά απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. Η 129 απορρίπτεται. Τροπολογία 130 του κυρίου Λούκα Χάρτονγκ. Η συγγήτρια είναι κατά. ποιο είναι υπέρ? κατά αποχές απορρίπτεται 131 της κυρίας Τρίπελ κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα ζητά περαιτέρω μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων. Είναι υπέρ εισηγήτρια. Αλλά φαίνεται ότι δεν αρέσει στο ΕΛΚΑ. Πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 24 ψήφοι συν 1, 25 υπέρ, 14 ψήφοι κατά, το πρώτο τμήμα εγκρίνεται κατά του ΕΛΚ. Δεύτερο τμήμα που είναι το υπόλοιπο. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Hey there. Uh c'est gentil, c'est sympathique, mais c'est minoritaire. Et donc... <laughs> Λοιπόν, το δεύτερο τμήμα επίσης εγκρίνεται. Και μέσω προφορικής τροπολογίας ε, θα ε, προσθεθεί στην παράγραφο 38. Και δεν θα έχουμε 38α νέα. Έχουμε περίπου 6 τροπολογίες που καταπίπτουν αυτές που ακολουθούν και πάμε στην 138 του κυρίου Χάρτονγκ. Η κυρία Σιγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 139 Μοργάντη. Σιγήτρια είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 140 Χάγκλοντ. Η Σιγήτρια είναι κατά. Υπέρ. 6 κατά οι περισσότεροι άποχες απορρίπτεται 141 Helga Triple, η συγγήτρια είναι υπέρ αλλά το έλκ είναι κατά ηλεκτρονικός έλεγχος 141 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 141 τέλος ψηφοφορίας «20 συν 21 ψήφι υπέρ, 18 κατά, μικρή διαφορά υπέρ, εγκρίνεται 141. Οι άλλες τροπολογίες καταπίπτουν μέχρι την 148 της κυρίας Ανδρέασεν. Ψηφίζουμε. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 149 της κυρίας Ανδρεάσεν. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. 4. Κατά. Η πλειοψηφία. Αποχές απορρίπτεται. Και αυτή 150 της Γκουε. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Η Γκουε και η πράσινη. Η κυρία Βέρτμαν κατά. Η πλειοψηφία. Αποχές απορρίπτεται. 151 μπόκρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 152 Χαρτόγκ. Η είναι κατά. Πίσουν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 153 μπόκρους. Η είναι κατά. Πίσουν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 154. Μου λένε ότι η συντάκτρια της 154 που είναι ανάμεσά μας ζήτησε το λόγο. Μπάρμπαρα, θέλετε να μιλήσετε για την 154, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να παρουσιάσω μια προφορική τροπολογία, όπου προστίθεται στο κείμενο της τροπολογίας το εξή. Το άρθρο 2, πριν από το slowdown, πριν από το illegal migration, και μετά προσθέτουμε whilst acknowledging ότι τα κάτι μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με το, με το νόμο της Ευρωπαϊκής Ενώσης και τονίζει την ανάγκη και μετά αυτό το κείμενο ενώνεται με το κείμενο το αρχικό της δικής μου τροπολογίας. Καταλάβατε όλοι. Έχει διανεμηθεί το κείμενο αυτό. Καλώς. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία που τροποποιήθηκε από την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αρκετή. Εννέα απόχειος. Εγκρίνεται με την προφορική τροπολογία. Τροπολογία 155 Helga Triple. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι. Α, ηλεκτρονική ψηφοφορία. για την τροπολογία 155 που ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. ...16 υπέρ, 23 ψήφοι κατά, απορρίπτεται. 156 πόρτας. Η συγκήτρια είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. 5 κατά οι περισσότεροι αποχές απορρίπτεται 157 του Θόδωρου Σκυλακάκη η συγκίτρια είναι υπέρ ελληνική ψήφος κατά 3, 5 αποχές 2 εγκρίνεται 158 το αντιπροέδρο Αλβάρο η συγκίτρια είναι κατά ποιος είναι υπέρ 8 κατά η πλειοψηφία αποχές απορρίπτεται 159 χάρτον και η 3 είναι κατά ποιος είναι υπέρ 3 κατά αποχές απορρίπτεται 160 μοργάντι η 3 είναι κατά ποιος είναι υπέρ 3 κατά άποχες απορρίπτεται 161 του κυρίου Χάρτονγκ υπέρ 2 κατά αποχές απορρίπτεται 162 Μιγγέλ Πόρτας και άλλων κατά τμήματα πρώτο τμήμα takes the view μέχρι European Strategy η είναι κατά ποιος είναι υπέρ η Γκουε κατά υπόλοιποι αποχές το πρώτο τμήμα απορρίπτεται δεύτερο τμήμα reiterates μέχρι citizenship. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. 163 Μιγγέλ Πόρτας. Η συγκήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ? Μία ψήφος κατά. Οι υπόλοιποι αποχές απορρίπτεται. 164 Λούκας Χάρτον και η συγκήτρια είναι κατά. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 Χάγκλουντ, εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 166 του κυρίου Μπόκρος και 167 του κυρίου Χάρτον και είναι ταυτόσιμη. συγγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Τέσσερις. Κατά. Οι περισσότεροι αποχές απορρίπτονται. 168 του κ. Χαγκλούν. Η είναι κατά. Υπέρ. Έξι. Κατά. Οι περισσότεροι. Αποχές απορρίπτεται. Πάμε συνεχεία στο κάτω με σελίδες 174 της Προέδρου Ιούτα Χάουγκ που εκπροσωπεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ κατά 5 αποχές 1 εγκρίνεται συγχαρητήρια στην κυρία Χάουγκ 175 Χέλκα Triple η είναι κατά ποιος είναι υπέρ 2, 3 7 κατά αποχές απορρίπτεται 176 του κυρίου Χάρτονγκ η είναι κατά ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 177 του κυρίου Λαβία η Α, ποιος είναι υπέρ μάλλον συγγνώμη λέει πρόεδρος κατά αποχές εγκρίνεται 178 του κυρίου Μπόκρος η είναι κατά ποιος είναι υπέρ τέσσερις κατά οι περισσότεροι αποχές απορρίπτεται 179 της Helga Trippel με προφορική τροπολογία που αφορά την παράγραφο τις παραγράφους μάλλον ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας αυτής που υποστηρίζεται από την εισηγήτρια κατά τρεις αποχές εγκρίνεται. Άρα θα η παράγραφος 28 αντικαθιστά, την 23 180 ματέρα υπέρ κατά τέσσερις αποχές 2 εγκρίνεται Δύο ταυτόσιμε τροπολογίε περί διαγραφή τη κυρία Άντρεσεν και του κυρίου Χάρτονγκ. Η συγγήτρια είναι κατά ποιο υπέρ. Κατά. Αποχές 181 και 182 απορρίπτονται. Τροπολογία 183 αποσύρεται. Πάμε λοιπόν στην 184 του κυρίου Χάρτονγκ. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Τέσσερις κατά. Οι περισσότεροι εποχές απορρίπτεται. 185 Μοργάντι. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Τέσσερις. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 186 του κυρίου Χάγκλουντ. Η συγκίτρια είναι κατά. Υπέρ. Α, συγγνώμη. Η συγκίτρια είναι κατά, αλλά το έλκυν υπέρ. Διέρεση στον μαμούθ λοιπόν. Περνάμε στον ηλεκτρονικό έλεγχο. Πού ξεκινά ο έλεγχος, η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ας βιαστούμε, ας βιαστούμε. Πέρας ψηφοφορίας. Τέλος 22 συν 1, 23 υπέρ. 15 κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία 187 του κυρίου Λαβία. Η συγγήτρια είναι υπέρ υπέρ κατά εννέα αποχές οι περισσότεροι είναι υπέρ εγκρίνονται η τροπολογία 188 Λούκας Χάρτον και η συγκέντρια είναι κατά ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 189 του κυρίου Μοργάντη η συγκίτρια είναι κατά ποιος είναι υπέρ 4 κατά οι περισσότεροι αποχές απορρίπτεται. 190 του κυρίου Χαγκλούν. Η συγκήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος εδώ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία όσον αφορά την 190 ξεκινάει η ψηφοφορία. Πολύ σιγά προχωράμε. Βιαστείτε λίγο. Είναι κάποιοι θέλουν να ψηφίσουν. Λοιπόν, πέρας. 17 υπέρ. 19 συν 1, 20 ψήφοι κατά, απορρίπτονται. 191, Μόνικα Όλμαερ. Η συγκήτρια είναι κατά. Υπέρ. 3, 4, 6, 7. Κατά. Οι περισσότεροι Όλη η ομάδα κατά της κυρίας Χολμάιερ αποχές. Η τροπολογία αυτή απορρίπτεται 192 του κυρίου Μοργκάν Η συγγήτρια είναι κατά ποιος είναι υπέρ της 192. Κατά αποχές απορρίπτεται 193 του κυρίου Χάρτονγκ. Η συγγήτρια είναι κατά ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 194 του κυρίου Χάρτονγκ εισηγείται είναι κατά ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 του κυρίου Χάρτονγκ εισηγείται είναι κατά ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 196 του κυρίου Χάγκλουντ εισηγήτρια είναι κατά ποιος είναι υπέρ 8 κατά. Αποχές απορρίπτεται. 197 της κυρίας Ανδρεάσης, εισηγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. 4 κατά. Αποχές απορρίπτεται. 198 του κυρίου Μποκρός. Εισηγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. 2 κατά. 3 μάλλον υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Απορρίπτεται. 199 της κυρίας Αντρεασέν, η συγγήτρια είναι υπέρ, ε, κατά συγγνώμη, ποιο είναι υπέρ. 4-5 κατά. απόχέ απορρίπτεται. 200 του κυρίου Φερνάντες, η συγγήτρια είναι υπέρ. Κατά. 3 Αποχέ, 2 εγκρίνεται. 201 της κυρίας εν συγγήτρια είναι κατά. Α, η 201 καταπίπτει διότι 200 εγκρίθηκε για την ίδια παράγραφο. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε στη 202 τη κυρία Ανδρεάσεν. Η συγγήτρια είναι κατά. ποιο είναι υπέρ? Τέσσερις κατά. Η πλειοψηφία αποχές απορρίπτεται. 203 του κυρίου Χάρτον. Η συγγήτρια είναι κατά. ποιο είναι υπέρ? Τέσσερις κατά. Αποχές απορρίπτεται. 204 του κυρίου Χάγκλον. Η συγγήτρια είναι, κατά... είναι ταυτόσιμη με τη 205 και τη 206. Τρεις τροπολογίες λοιπόν για την ίδια ψήφο. Ποιος είναι υπέρ. 13 Κατά. Σηκώστε τα χέρια. Καλά να είμαστε σίγουροι. Πλειοψηφία λοιπόν, αποχές, αυτές οι τρεις τροπολογίες απορρίπτονται. 207 του κυρίου Λαβία, εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Όλοι οι σοσιαλιστές είναι κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν. Ζητώ συγγνώμη. Νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία, αλλά να επαληθεύσουμε. 207 του κυρίου Λαβία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας 26 συν 1, 27 ψήφοι υπέρ, 11 κατά, οι είναι απομονωμένοι στην εχθρική του στάση. Λοιπόν, 207 εγκρίνεται, 208, 208 ε, καταπίπτει. Πάμε σε 209 και 210 που είναι ταυτόσημες, η συγγήτρια είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Τέσσερις ψήφοι κατά, οι περισσότεροι αποχές απορρίπτονται. 211 του κ. Μπόκρος. Η είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. 4. Η ύποπτη. Συν τον Τζέιμς Έλλες... 5. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 212 του κ. Χάγκριν. Η είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Επτά κατά αποχές απορρίπτεται. 213. Άστριγκ Λούλινγκ της πρεσβυτέρας μας. Ε, είναι υπέρ προφανώς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Η 213 εγκρίνεται. 214 του κυρίου Λαβία η συγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 215 του κυρίου Λαβία σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα underlines that μέχρι key services η συγγήτρια είναι υπέρ ποιος είναι υπέρ κατά άποχες το πρώτο τρίτο τμήμα μέχρι has been applied. so Steve μέχρι has been applied. Η συγγήτρια είναι κατά αυτή τη φορά. Λοιπόν, Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της 215. Άρχεται η ψηφοφορία. Προχωράει αργά η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. Λοιπόν, 15 ψήφοι υπέρ, 22 συν 1 ψήφος, 23 ψήφοι κατά. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. 216 της κυρίας Άντρες, ενισχύτρια είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 217 του κυρίου Λαβίας, η γητρία είναι υπέρ, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία για την παράγραφο 71 της Φραντσέσκα. Την έχετε μπροστά σας. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά Αποχές. Η προφορική τροπολογία εγκρίνεται. 218 του κυρίου Μπόκρος. Η είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Έξι κατά. Η περισσότερη απορρίπτεται. 2.19 του κυρίου Χάρτονγκ. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 220 του κυρίου Μοργκάντ τι είναι κατά η συγκήτρια, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 221 Μάρτα Άντρεσαν η συγκήτρια είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 222 του Λούκας Χάρτον και η συγκήτρια είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 223 της κυρίας είναι συγγήτρια. είναι κατά. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 224 της κυρίας Η συγγήτρια. είναι κατά. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Είναι ταυτόση με 225 που και αυτή απορρίπτεται. 226 του κυρίου Χάρτονγκ συγγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά Αποχέ, απορρίπτεται 227 της κυρίας Ανδρεάσεν συγγήτρια είναι κατά ποιος είναι υπέρ κατά Αποχέ, απορρίπτεται 228 του κυρίου Χάρντον και συγγήτρια είναι κατά Ποιο είναι υπέρ κατά Αποχέ, απορρίπτεται 229 του κυρίου Μοργκάντη συγγήτρια είναι κατά ποιος είναι υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 230 Γιούτα Χάουκ, εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Τρεις αποχές εγκρίνεται. 231 καταπίπτει διότι εγκρίναμε την τροπολογία 82. η Γιούτα μπορεί να θεωρήσει ότι καλύπτεται ήδη η τροπολογία της, η, η τροπολογία του 31. 232, Χάρτονγκ, η συγκήτρια είναι κατά, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 233 του κυρίου Χάγκλουντ, η συγκήτρια είναι κατά, Ποιο είναι υπέρ, Επτά κατά. Οι περισσότεροι αποχές απορρίπτεται. 234 Γιούτα Χάουγκ. Η συγκέντρια είναι υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.35 του κυρίου Χάρτονγκ, η συγκέντρια είναι κατά, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.36 της κυρίας Γιούτα η συγκέντρια είναι υπέρ, υπέρ, κατά, τέσσερις αποχές εγκρίνεται 237 καλύπτεται πάμε στην τροπολογία 1 είμαστε λοιπόν στις αναφορές εδώ ε, τροπολογία 1 εν ονόματι της Επιτροπής ΕΜΚΟ δεν θέλει η συγγήτρια είναι κατά είναι υπέρ λοιπόν... ηλεκτρονικός έλεγχος της ψηφοφορίας για την ε, υπαριθμόν 1. άρχιτε ψηφοφορία. Πέρασε. 17 υπέρ, 20 και 1 κατά, απορρίπτεται. 2. James Ellis. Συγγήτρια είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. 6. Κατά. Πλειοψηφία. Αποχέ. Απορρίπτεται. 3. James Ellis. Ζηγείται είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Η ίδια πλειοψηφία. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές απορρίπτεται επίσης. Τέσσερα. Κυρία Θαμπάλ. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Δύο συνάδελφοι δεν ψηφίζουν. Λοιπόν, 20 σημεία, 21 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται η τροπολογία. 5. James Ellis, εσύ γιατί είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Πλειοψηφία. αποχέ. Απορρίπτεται. 6. James Ellis. Υπέρ. Κατά. Η ίδια πλειοψηφία. Απορρίπτεται. Λοιπόν, η γραμματεία μου λέει ότι λόγω τρόπου με τον οποίο εργαστήκαμε χάρη στην και του συντονιστέ μα και δεδομένου ότι οι κύριε γνωμοδοτήσεις των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών ρίχνει υπόψη από τις τροπολογίες ή και απορρίφθησαν από τις τροπολογίε, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε κάθε μία από τις γνωμοδοτήσεις αυτές των επιμέρους κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θα τι παρατήσουμε στην ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία λοιπόν. Α, συγγνώμη, James. Συνήθως στην παρά... περίπτωση αυτή υπάρχει μια παράγραφο στο ψήφισμα που λέει ακριβώς ότι καλύπθηκαν οι απόψει των άλλων επιτροπών, αλλά θα έχουμε διαμαρτυρίες. Ναι, ευχαριστώ James που ε, δικαίως μας ε, υπενθύμησε στην παράδοση αυτή και θα υπάρχει αυτή η παράγραφο που αναφέρεται στον κατάλογο ψηφοφορία που έχετε μπροστά σα ούτω ή άλλω. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία. Στην ούτω τροποποιηθήσα έκθεση ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία έρχεται. Πέρας. Κύριε Πορτός, υπέρ τελική ψηφοφορία. Λοιπόν, 25 υπέρ, 7 κατά και 6 εποχές. Ωραία. Συγχαρητήρια στην εισηγητριά μας. Ευχαριστώ τους πάντες. Non, voter. Non, non. Euh, oui, mais bon, là, il y a discussion. Est-ce que c'est pas mieux de liquider les votes simples avant Alors, je vous propose de voter. Les Λοιπόν, προτείνω στο τέλος της πληροφορίας να ψηφίσουμε τους διορθωτικούς προεπιλογισμούς 2 και 3 που θα απαιτήσουν κάποια συζήτηση. Μπορούμε λοιπόν τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία για το σύστημα ευρωπαϊκών σχολείων. Έκθεση Σταμιέ Αμπάτ. Παίρνετε λοιπόν την λίστα ψηφοφορία για την έκθεση Αμπάντ. Είσαστε όλοι έτοιμοι. Tout le monde est prêt. Ne partez pas, Barbara. Nous votons. φύγετε, Μπαρμπαρά. Θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, ε, ψηφορία πάνω στην του κ. Αμπά. Τροπολογία 1, Αλβάρο. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Μια κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Καταπίπτει. Γιατί εγκρίθηκε η 1. Το ίδιο ισχύει για την 3. Περνάμε στην τροπολογία 4. Συντονία. Ο Εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Ε, Μια ψήφος κατά. Αποχές. Γκρίνεται. 5. Λούκα Χάρτο. Συγητή είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 6. Ο είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 7. Αλβαρό. Είναι συμβατή με την έκτη. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Εγκρίνεται. Οκτώ. Καταλήν Σολήν Ιβάν. Συγχτής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Για να ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 8. Είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Πέρας. 12 υπέρ, 23 και 1, 24 κατά. Η 8 καταπίπτει λοιπόν. Απορρίπτεται μάλλον. Η 9 χάρτου πρέπει να ψηφιστεί. Ψηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Δέκα, Αλβαρό. Ο ψηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Πέντε. κατά. Εποχές. εγκρίνεται. Έντεκα. Ο ψηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. ηλεκτρονικό και ψηφοφορία για την 11. Παρακαλώ. Oui. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Δεκαπέντε υπέρ, 22 κατά. Η 11 απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 12. Χάρτον. Προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχει το κείμενο. Κύριε Αμπά. Η, επόμενη είναι προφορική κύριε Πρόεδρε. Εδώ υπάρχει ένα ασφανο. Λοιπόν, η 12. Ψηφίζουμε τη 12. Χωρί προφορική τροπολογία. Συγχωρείτε είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Μία ψήφος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Ψηφίζουμε από αυτές επίσης. Α, εκεί υπάρχει η προφορική τροπολογία. Ναι, πράγματι, εκεί υπάρχει μια ψηφο υπερ τροπολογία, πρόεδρε. Και όπως φαίνεται, είναι η ίδια που έχετε. Αλλά θα διαγράψουμε την τελευταία μισή πρόταση ε, της παραγράφου 3 δηλαδή budget autonomy for schools. Η μουσιονομική αυτονομία για τα σχολεία. Έχετε όλο το κείμενο αυτό. Και υπάρχει ο στόχος να διαγραφεί το τελευταίο τμήμα τη πρόταση. Να σταματήσουμε δηλαδή εκεί που λέει το κείμενο Buildings Policy. Πολιτική κτηρία. Ωραία. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία αυτή που προτείνει ο εισηγητή. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Το στηρίζει ο συγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 14. 15. Ματέρα. Ο συγητής είναι κατά. Α, όχι. Είμαι υπέρ άλλαξε άποψη φαίνεται ο Κισίδης μετά από συνομιλία με την κυρία Ματέρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Για να μετρήσουμε. Αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία αυτή. Η 16 χάρτο. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική παρακαλώ. Άρχιε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα. 35 υπέρ, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Προτείνω να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία των δύο εκθέσεων της Προέδρου Γιούτα Χάουκ. Καταρχήν, σε εκείνη που προβλέπει εσύ σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Θα πρέπει να πάμε γλυβέρα μου φαίνεται. Γιατί η Γιούτα Χάουκ εργάζεται πάντα πολύ αποτελεσματικά. Σας προτείνει λοιπόν να ψηφιστούν on block οι τροπολογίες 1 έως 15. Ποιος είναι υπέρ του μπλοκ αυτού των τροπολογιών. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Δεκαπέντε τροπολογίες, 1 15 εγκρίθηκαν. Τελική ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ίδια πλειοψηφία. Ομοφωνία. Εκτός από την κυρία Ανδρεάσεν. Περνάμε τώρα στη δεύτερη έκταση Γιούτα Χαόκ για την... τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, την ΕΝΙΣΑ οποίο πάλι έχουμε ένα μπλοκ που καλύπτει τις τροπολογίες 1 έως 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Εγκρίνονται. Τροπολογία 17. Καλφίν. Με μια προφορική τροπολογία που έχετε μπροστά σας. που προσθέτει comprehensive analysis, related elaboration κλπ. κλπ. Οπωσδήποτε η εισήγητρια δεν τη θέλει η επιλογή αυτή. Άλλαξα γνώμη, λέει η κυρία Χάουγκ. Και εσείς μετά από προσωπική συνομιλία με τον υποβάλλοντα. Όχι προσωπική, λέει η κυρία Χάουκ, με email έγινε επικοινωνία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τροπολογία 17. Με προφέρει και τροπολογία. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Τροκαλύπτει την 10 Περνάμε τώρα στη 18 του κυρίου Αλβαρό. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ? 10, 11, 12. Ποιος είναι κατά? Κατά παρακαλώ. Αμπαχές. Απορρίπτεται. 19 του κυρίου Αλβάρο. Υπέρ. Η ίδια της πλειοψηφίας νομίζω. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. Φαντάζομαι θα είναι ικανοποιημένος ο κ. Σαλβάρο από αυτή την σύντομη ήττα. Τέλο πάντων. Κάλυψαν 13. 14 κάλυψαν. για την υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 15 Αλβαρό. Υποστηρίζει η συγκεντρή. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Μπαλτσίτης. Με μια προφορική τροπολογία. Να διαγραφεί η λέξη more, περισσότερη διαφάνεια. Να έχουμε διαφάνεια δηλαδή, όχι και υπερβολικά πολύ. Λοιπόν, με αυτή την προφορική τροπολογία που είναι υπέρ, η συγκέντρα ποιος είναι υπέρ. Κατά. Σε αποχές Σαρπάσια Συγχαίρουμε τον Παπαδάλη για την τροπολογία τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 34 υπέρ, μία κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια Γιούτα. Τώρα, μπορούμε νομίζω να περάσουμε τις ψηφοφορίες των εκθέσεων της Ιδονίας. Εσείς τώρα. Ce que je vous propose peut-être, c'est que vous nous présentiez θα έλεγα να μας προτείνετε τις προτάσεις για το διορθωτικό του προπορισμού 2 και 3, γιατί υπάρχουν πολιτικός συσχετισμός μεταξύ των δύο. Θα έχουμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων και μετά αν θέλετε μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία ή θα αναβάλουμε την ψηφοφορία. Συνδονία. έχετε τα λόγο. Νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε την έκθεσή μου για την, τον δεύτερο τροποποιητικό προπολογισμό συμπεριλαμβανομένη και, της προφορι... και, και των προφορικών τροπολογιών. Δεν ξέρω αν τι έχετε πάρει τις τροπολογίες μου. Ε, ας συζητήσουμε τον τρίτο διορθωτικό σήμερα, αν συμφωνείτε. Εσείς θα αποφασίσετε αν θα τα συνενώσουμε. Κατά την άποψή μου μπορούμε να τα χωρίσουμε γιατί τον δεύτερο διορθωτικό το συζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίασή μας. Σας διένυμα, μάλλον σας έστειλα με email της, προ, μου, ίσως θα έπρεπε να σας εξηγήσω το σκεπτικό τους. Ε, ακολουθούν την δήλωση της ε, Κομισιόν ε, που σχετίζεται με την ε, υπό εφαρμογή ενός από, τους, ενός από τα προγράμματα και στις 17 Ιουνίου αν θυμάστε πήρατε και εσείς και εγώ μια επιστολή από τον Επιτρόπο Λεβαντόφσκι την οποία εγώ ερμηνεύω ως αλλαγή του αρχικού του προσχεδίου τροποποιητικού προϋπολογισμού. Εκεί, σε αυτήν την επιστολή, προτείνει ε, το ποσό το οποίο είναι απαραίτητο για την κινητοποίηση του ε, Ταμείου Λεγγύης. Ε, λαμβάνω υπόψη και αυτή την επιστολή λοιπόν στην ε, προφορική μου τροπολογία και είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν διαφωνίες η δική μου ερμηνεία ε, σχετίζεται με τον τρίτο διορθωτικό ε, προϋπολογισμό. Ε, νομίζω όμως ότι μπορούμε να ψηφίσουμε τον δύο. Bien, je vous remercie. Euh, Anne Jensen. Yes, thank you, Έγιναν συζητήσεις για, εκεί για το δεύτερο και για τον τρίτο διορθωτικό προπολογισμό. Τα χρήματα για τον δεύτερο διορθωτικό προπολογισμό κατόπιν ε, πρόταση στη Συντόνια προέρχονται από μη δαπανηθέντα ποσά ε, ενεργειακών προγραμμάτων. Τώρα είναι λίγο νωρί για να πούμε ότι ε, αυτό το α ή το β δεν πρόκειται να ε, χρησιμοποιηθεί κλπ. Αλλά η Κομισιόν μας ενημέρωσε ότι ορισμένα από τα ενεργειακά project του σχεδίου ανάκτηση δεν θα πραγματοποιηθούν, δεν θα υλοποιηθούν ή μάλλον θα υλοποιηθούν με καθυστερήσει, οπότε αυτά τα χρήματα, αυτά τα κονδύλια θα είναι διαθέσιμα για το 2011, εξού και η μεταφορά μέσω του διορθωτικού προπολογισμού. Αυτές ήταν οι πληροφορίες που είχαμε όταν τελευταία συζητήσαμε τον τρίτο διορθωτικό προπολογισμό όπου συζητούσαμε να, τα χρήματα να προέρθουν από το πλεόνασμα του περασμένου έτους και εξετάσαμε το κατά πόσο αυτό είναι δυνατό. Εγώ εκ μέρους ομάδας μου είχα ένα αντίθετο επιχείρημα να γνωρίζω ότι δεν εξασφαλίζουμε πλειοψηφία αλλά από ό,τι κατάλαβα είχαμε ζητήσει και από την νομική υπηρεσία να μας πει ποια θα ήταν, ποια, αν υπάρχει δυνατότητα να υποβάλουμε τον τρίτο διορθωτικό προπολογισμό υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν άκουσα ακόμα την απάντηση των νομικών υπηρεσιών. Ε, νομίζω ότι θα ήταν ε, χρήσιμο, τουλάχιστον από τη δική μας ομάδα, αυτό πιστεύουμε, θα ήταν χρήσιμο να την ακούσουμε. Σαλβαδόρ και εμείς το συζητήσαμε στην ομάδα μας. Συζητήσαμε και, τα δύο, και τους δύο διορθωτικούς προπολογισμούς και συμφωνούμε με την Σιδόνια που προτείνει να γεμίσουμε το συντομότερο δυνατό την, το αρνητικό απόθεμα που είχαμε δημιουργήσει. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε κάποια στοιχεία για την εκτέλεση του προπολογισμού που δείχνουν ότι υπάρχει μια υστέρηση στην εκτέλεση. Είναι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα στον δεύτερο διορθωτικό προπολογισμό για μια σειρά από πολύ σαφείς στόχους. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο διορθωτικό προπολογισμό, περιμέναμε ακόμα περιμένουμε την <laughs> άποψη τη νομική υπηρεσία, αλλά από, ότι, από τις προφορίες που έχουμε πάρει οι συντονιστές φαίνεται πως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πραγματική δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με το Συμβούλιο σε αυτή τη στιγμή της δημοσιονομικής διαδικασίας. Δηλαδή να τροποποιήσουμε ένα ε, προπολογισμό ε, ε, περισσευμάτων είναι κάτι πολύ πιο λογικό. Δεν νομίζω ότι τον Ιούνιο θα έπρεπε να είναι δυνατόν να συζητηθεί αυτό το ζήτημα. Ίσως όταν συζητηθούν οι επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές ή σε κάποια, κάποια στιγμή αργότερα τουλάχιστον ε, αυτό το χρόνο νομίζω ότι αυτή τη στιγμή καλύτερα να ακολουθήσουμε την πρόταση τη συντόνια ε, με τον δύο τροποποιημένο και τον τρία χωρίς καμία τροποποίηση. Ευχαριστώ ο κ. Μπόκρος. Because ψηφίσαμε εναντίον της ε, απλοποίησης και υπέρ του reshuffle, της αναδιανομής, ανακατανομής. Αυτό είναι, αυτή είναι μια πραγματική ανακατανομή στο πλαίσιο του υπερπολισμού του 2011 και νομίζω ότι ε, είναι κακή επιλογή, αλλά οι άλλες είναι ακόμα χειρότερες επιλογές. Συνεπώς θα ήθελα να ψηφίσουμε υπέρ. Γιατί το χειρότερο, το χείριστο θα ήταν να διατηρήσουμε το αρνητικό απόθεμα. Συνεπώ, αν η Κομισιόν λέει ότι αυτό είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε, ε, ε, δεν είναι πολύ κομψή η λύση, αλλά καλύτερο από το να διατηρήσουμε ε, αιωνίω το αρνητικό απόθεμα. Γκόραν Φέρμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Συμφωνώ πλήρω με του προηγούμενου ομιλητέ στον ε, διαρθρωτικό προϋπλασμό υπαριθμών 2 είμαστε υπέρ της ε, διόρθωσης που πρότεινε της τροπολογίας πρότεινε η συγγήτρια το, η θέση του Συμβουλίου είναι να αρνηθεί ε, οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη λύση εκτός από αυτήν προτείνει το ίδιο είναι λάθος αυτή η στάση σε ό,τι αφορά τον τρίτο διορθωτικό προπολογισμό θα ήταν ενδιαφέρον να το δοκιμάσουμε αλλά μάλλον για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο όχι για αυτό όπως είπε και ο Σαλβαδόρ νομικά θα είχαμε πολύ συχνά επιχειρήματα να αρνηθούμε αυτό τον προπολογισμό, οπότε συμφωνούμε με την εισηγήτρια. Ευχαριστούμε, Γκέρεν, Πολύ σαφές το, το, αυτό που είπες. Κυρία Ματέρα. Θα είμαι πολύ σύντομη, λέει η κυρία Ματέρα. Θέλω να υποστηρίξω πλήρω την πρόταση τη Συντόνια όσον αφορά τη μεταφορά των χρημάτων που δεν χρησιμοποιήθηκαν και ανήκουν στη γραμμή του προπολογισμού ενεργειακά προγράμματα είναι υποστήριξη τη οικονομική ανάκαμψη υπέρ του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Μιλάω σαν standing, μόνιμη συγγήτρια για το Ταμείο αυτό τη προσαρμογή στην ε, ε, παγκοσμιοποίηση. Πλήρη υποστήριξη προ την συντόνια. Ευχαριστώ. Η συντόνια θα μας προτείνει μια λύση έχοντας ακούσει τις απόψεις όλων εγώ προτείνω το εξή. Θα ψηφίσουμε για τον δεύτερο διορθωτικό προπολογισμό με τις τροπολογίες που μας προτείνει η συγκήτρια. Τώρα, θα γίνει ψηφοφορία τώρα, όπω το είχαμε προβλέψει. Είχαμε επίση προβλέψει ότι ο τρίτος διορθωτικός προπολογισμό θα ψηφιστεί στην επόμενη συνεδρίασή μας. Συνεπώ, προτείνω, αν είναι να ψηφίσουμε τον δεύτερο διορθωτικό, μετά την ψηφοφορία, για να προετοιμάσουμε την άποψή μας για τον τρίτο διορθωτικό προπολογισμό, θα δώσω το λόγο στην νομική υπηρεσία για να μας παρουσιάσει προφορικά την ανάλυση της για τα νομικά προβλήματα τα οποία δημιουργεί ο τρίτος διορθωτικός προπολογισμό. Θα μας στείλει την γραπτή της αναφορά αργότερα. Αλλά μια προφορική παρουσίαση θα μας επιτρέψει ε, να τοποθετηθούμε και να προετοιμάσουμε την ψηφοφορία για τον τρίτο διορθωτικό προπολογισμό. Κυρία Σίγητρε, ο λόγος εσά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους ομιλητέ, να ευχαριστήσω όσους με υποστήριξαν. Δεν λέω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση, είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Λάβατε την έγγραφο με τις τροπολογίες μου. Καλύτερα θα ήταν, Πρόεδρε, να τις εξηγήσω λιγάκι. Η ιδέα είναι η εξή. Αναφέρθηκα στην επιστολή της Κομισιόν, η οποία μιλάει μόνο για τα 19 εκατομμύρια για το Ταμείο Ελεγγύης, τις πληρωμές του Ταμείου Ελεγγύης. μου οι δικές μου τροπολογίες όμως πάνε πιο μακριά. Σε κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στην επιστολή της Κομισιόν. Έχουν ως στόχο να εξορροπηθεί, να μικρυνιστεί το αρνητικό απόθεμα και όπως είπε η Μπάρμπερα, να προσθέσουμε κονδύλια για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Πώ έχουμε δύο επιπλέον στοιχεία. Ε, αυτή η τροπολογία θα δημιουργήσει ε, σύγκρουση με το Συμβούλιο. Αυτό το λέω για όσους είναι συγκρουσιακοί για σχέση με το Συμβούλιο. Ε, δεν είναι τόσο απαλές αυτές οι τροπολογίες, ούτε ανώδυνε, γιατί ε, με αυτές τις τροπολογίες ε, αν, μάλλον αν αυτές οι τροπολογίες συγκριθούν η, το Συμβούλιο θα τις ερμηνεύσει ως επιθετική κίνηση, γιατί το Συμβούλιο και οι Κομισιόν περιμένουν από εμά να περιμένουμε ευγενικά μέχρι να έρθουν τα αιτήματα για μεταφορές. Επειδή όμως βλέπουμε προβλήματα, επειδή εγώ βλέπω ότι το αρνητικό απόθεμα είναι εκρεμέ ζήτημα και θα πρέπει να λάβουμε πρωτοβουλία να το ρυθμίσουμε. Γι' αυτό προτείνω αυτέ τι τροπολογίε με τρία στοιχεία. Δεν ξέρω αν θα μα οδηγήσουν σε συνδιαλλαγή. Ελπίζω όχι. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα είναι αρκετά έξυπνο για να δει την καλή μας πρόθεση και να, και να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν δύο ακόμα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν, το αρνητικό απόθεμα και το, το της του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα δείξει εξίσου καλή πρόθεση, ε, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε. Ωραία. Νομίζω ότι όλα είναι πολύ σαφή. Έχουμε μια ευρεία συνένεση, όχι ομοφωνία, αλλά συνένεση. Είμαστε πίσω, υποστηρίζουμε την συγκήτριά μας. Ε, στο ΚΑΠΑ, στο συμβασμό ΚΑΠΑ, ας προσθέσουμε τον κατάλογο των βασικών θεμάτων τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στον τριμερή διάλογο της 11 η Ιουλίου λέγοντας ε, τα προβλήματα, τα εκκρεμή προβλήματα του προπολισμού, της εκτέλεσης του προπολισμού του 2011 ε, θα πρέπει να αναφερθούν, να συζητηθούν στις 11 Ιουλίου, να πούμε κάτι τέτοιο. Δεν επιθυμούμε σύγκρουση με το Συμβούλιο, αλλά αναφέρουμε με σαφήνεια ότι δεν έχουμε την ίδια προσέγγιση με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά ε, τα, τις απρόβλεπτες ε, δαπάνες ε, τις μη προβλέψιμες δαπάνες του 2011, ούτε καν ερμηνεύουμε με τον ίδιο τρόπο την δήλωση που υιοθετήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο ως παράρτημα της συμφωνίας μας για τον προπολογισμό του 2011, δήλωση σύμφωνα με την οποία οι απρόβλεπτες δαπάνες του 2011 θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν ε, με πρόσθετους πόρους ε, ως πιστός πληρωμών. Λοιπόν, Πάρτε τον κατάλογο ψηφοφορία ε, για τον ε, διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 2. Θα ψηφίσουμε τις δημοσιονομικές τροπολογίες πρώτες, ενδεχομένως όλες μαζί, ομαδοποιημένες, όπως κάνουν προηγουμένως με τις τροπολογίες Χάουκ. Ε, οι τέσσερις τροπολογίες, δημοσιονομικές τροπολογίες, ποιος είναι υπέρ, όλες μαζί. Κατά. Αποχές καμία αποχή, υιοθετούνται. Τροπολογίες στο ψήφισμα τώρα. Μπορούμε και αυτές να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και μια προφορική τροπολογία την οποία έχετε μπροστά σας. Το Restoring Draft Amendment κλπ. αντικαθίσταται από το Covering the Needs Showing from the Mobilization ε, τι ανάγκε ανάγκες ε, από την κινητοποίηση του Ταμείου. Ε, ποιο είναι υπέρ, ποιο είναι κατά όλων αυτών των τροπολογιών. Αποχές εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Ομοφωνία μείον ένα. Δεν χρειάζεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ευχαριστούμε Συντόνια. Έκθεση Μπέργκε για το ίδιο θέμα, μια και είμαστε εδώ. Και μετά θα δώσω το λόγο στην νομική υπηρεσία. Έκθεση Ράιμερ Μπέργκε. Μία μόνο τροπολογία του κ. Χάρτογκ. Ο εισηγητής διαφωνεί. Ποιος είναι υπέρ. Μία ψήφος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ της έκθεσης Ράια Μερμπέγκε, κατά, μία ψήφος κατά. Κύριε Σουριάν, αποχές, εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. Τώρα, Στρέφομαι προς τον ε, Διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε την ανάλυση σας για δύο θέματα τα οποία συνδέονται σε πολιτικό επίπεδο και είναι τα εξή. Πρώτον, τι περιθώριο ελιγμών διαθέτει το Κοινοβούλιο Αναφορικά με την ε, χρήση πλεονασμάτων της προηγου, του προηγούμενου έτους, χρήση η οποία θα μπορούσε να γίνει μέσω ενός διορθωτικού προπολογισμού των υπαριθμών 3 φέτος, που όμως ε, προφανώς δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο διορθωτικό προπολογισμό. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση Σε ό,τι αφορά τα έσοδα του ευρωπαϊκού προπολογισμού, μπορούμε από νομικής πλευράς να θεωρήσουμε ότι στους υπολογισμούς του, των πλεονασμάτων εκτέλεσης, τα έσοδα τα οποία προέρχονται από πρόστιμα που έχουν πληρωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν αποφάσεων της Κομισιόν μπορούν να μπορούμε να τα μεταχειριστούμε με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που έχουμε και στην Επιτροπή και στην ομάδα των, των συντονιστών. Χρειαζόμαστε διευκρινήσεις από τη δική σας πλευρά για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε επί του διορθωτικού Περθυμοντρία. 3. Κύριε Διευθυντά. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα απαντήσω μία προς μία τις ερωτήσεις. Ό,τι αφορά τον διορθωτικό προπολογισμό υπαρτιμών 3, όπως είπατε και εσείς ο ίδιος ε, πρόεδρε, πρόκειται για έναν ιδιαίτερο διορθωτικό προπολογισμό που υποβλήθηκε από την Κομισιόν επί τη βάση του άρθρου 15 παράγραφος 3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Σύμφωνα με αυτή την διάταξη, μετά την παρουσίαση των λογαριασμών κάθε έτους, οποιαδήποτε διαφορά από τις εκτιμήσεις θα εντάσσεται στον προπολογισμό του επόμενου έτους μέσω ενός διορθωτικού προπολογισμού που ε, θα αφιερώνεται αποκλειστικά για τη ρύθμιση του συγκεκριμένου ζητήματος. Οπότε το, το μόνο αντικείμενο αυτού του διορθωτικού προπολογισμού είναι η χρήση του πλεονάσματος από το προηγούμενο έτος. Αυτή η διάταξη του άρθρου 15 παράγραφος 3 αναφέρει, όπως είπαμε, ότι αυτό Τόσο ο προϋπολογισμός, ο δοθετικός, αφορά, αφιερώνεται μόνο σε αυτό το ζήτημα και ε, αυτό καθιστά ε, τον προπολογισμό τεχνικής φύσης, τη, διορθω, τη διόρθωση τεχνικής φύσης και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να τη δεχτεί όσο έχει χωρίς τροπολογία, χωρίς τροποποίηση. Ε, αυτό προκύπτει από τη δική μας ερμηνεία του άρθρου 15 παράγραφος 3 που λέει ότι θα αφιερώνεται αποκλειστικά κλπ. κλπ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εισάγουμε άλλα ζητήματα. Αυτή είναι η απάντησή μου λοιπόν στο, στην πρώτη σας ερώτηση. Στη δεύτερη ερώτηση τώρα. Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα και το, και το κατά πόσον θα ε, μπορούσαν να τύχουν ιδιαίτερη μετα, ε, και να μην επιστραφούν στα κράτη-μέλη. Το θέμα αυτό είναι πολιτικής ε, φύσεως, άπτεται της πολιτικής σφαίρας. Οπότε εγώ απλώς θα προσπαθήσω να φερθώ μόνο στη νομική του πτυχή ε, και μπορώ να πω μόνο το εξή. Το άρθρο 15 του Δημοσιονομικού Κανονισμού έχει ως στόχο να εφαρμόσει την αρχή της ισορροπίας, της ε, ισοσκέλησης του προπολογισμού. Αυτό άλλωστε είναι και ο τίτλος του, άρθρου, του κεφαλαίου 3, στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 15. Αυτή η αρχή σημαίνει ότι τα έσοδα και οι δαπάνες ε, θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα. Το οποίο σημαίνει ε, ότι ε, τα πρόστιμα του, του ανταγωνισμού αποτελούν τμήμα των εσόδων. Αν θέλουμε να επιχειρηματολογήσουμε ότι τα πρόστιμα αυτά δεν πρέπει να επιστραφούν στα κράτη-μέλη, Πιστεύουμε ότι αυτό το επιχείρημα δεν θα ε, κάνει, δεν, θα, δεν σέβεται, ε, δεν συμμορφώνεται με την αρχή του ισοσκελισμού του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εξηγήσεις τις αφέστατες. Αν θα είχατε την καλοσύνη γραπτός να μας το υποβάλλετε αυτό <clears throat> το ώστε όλοι να μπορούμε εδώ να έχουμε την ενημέρωση με αυτές εβδομάδες, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Κυρία Συγήτρια, έχετε άλλες ερωτήσεις να θέσετε στην νομική υπηρεσία. Όχι. Ωραία. Πολύ καλά. Καλώς. Προτείνω να σταματήσουμε εκεί όσον αφορά την ψηφοφορία του διορθωτικού προπολογισμού. Θα ψηφίσουμε τον προπολογισμό υπαριθμών 3 την επόμενη εβδομάδα. Στην επόμενη συνάντηση, 27 το μηνό. Το χρονοδιάγραμμα μα υποχρεώνει μα το κάνουμε αυτό. Διότι αν δεν ψηφίσουμε, την τελευταία η τελευταία ευκαιρία θα είναι νομικά η Ολομέλεια του Ιουλίου, αυτό θα σήμαινε ότι η σιωπή σημαίνει συνένεση και το ότι το Κοινοβούλιο δεν υιοθέτησε καμία τροπολογία εντός των προβλεπωμένων προθεσμιών, προβλεπωμένων από τις συνθήκες για ένα σχέδιο διευθυντικού προπολογισμού, αυτό σημαίνει ότι συμφωνεί απόλυτα το Κοινοβούλιο με την ψηφοφορία του Συμβουλίου. Ε, και προφανώς δεν είναι αυτό που θέλουμε. Θα πρέπει λοιπόν να ε, ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών το διθωτικό προπολογισμό 3 κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδριάσεως μας 27 του μηνός. Αντίθετα έχουμε κάποιες ψηφοφορίες ακόμα και κυρίως μεταφορές έχουμε να κάνουμε. Όσον αφορά το διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 3, η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 20 Ιουνίου ε, το μεσημέρι. 12 το μεσημέρι. Θα πάμε τώρα στην, ε, στη ψηφοφορία των μεταφορών. Λοιπόν, κατηγορία 3. Θα δώσω ξανά το λόγο στη Συντόνια που έχει κάποιες μεταφορές να μας ε, προτείνει. Συντονιά. Vous avez ντρέπομαι, πώς να το πω, δεν έχω τον κατάλογο των μεταφορών, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε μια σημαντική μεταφορά που σχεδια... σχετίζεται το ΣΥΣ 2 και είναι η μόνη επίμαχη μεταφορά που έχουμε σήμερα, η δύσκολη και αν επιτρέπετε θα ήθελα να αναφερθώ στο ιστορικό και στη θέση μου. Δηλαδή υπήρχαν προβλήματα με την εφαρμογή του προγράμματος ε, ΣΥΣ και εγώ και η Μόνικα Χολμάιερ, ο κύριος Αλβάρου προσπαθήσαμε να ελέγξουμε το πώς το πρόγραμμα ΣΥΣ 2 εφαρμόζεται και στην ε, διαδικασία του προπολογισμού βάλαμε ένα αποθεματικό ε, θα μπορούσα να προσπαθήσω να εξηγήσω. Προσπαθήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσουμε για να μάθουμε περισσότερα. Τελικά τι μας είπαν. Ε, μας δώσαν αρκετές εξηγήσει κατά την άποψή μου για να μπορέσουμε εμείς να εγκρίνουμε τη μεταφορά εκτός αν οι συνάδελφοί μου που επίσης επεξεργάζονται το θέμα έχουν αντίρρηση θα έλεγα να ε, ψηφίσουμε υπέρ. Πολύ καλά. Είμαστε στη μεταφορά υπαριθμών 18, έτσι και είναι ένα θέμα που ήδη συζητήσαμε, το πρόβλημα του αποθεματικού για το σύστημα SIS-2. Μόνικα, ε, έχεις κάποιο σχόλιο? Θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω αυτά που είπε η Σιδρόνια. Ότι είχαμε μια τεχνική συνάντηση με την Κομισιόν και η Κομισιόν εκεί μας είπε αναλυτικά γιατί χρειάζεται αυτό, ποιο είναι το συμπληρωματικό κόστος, γιατί ήδη στις αρχές του, του ήταν σαφές ότι το κόστος θα ξεπεράσει το προπολογισμό, δεν ήξερα ακόμα κατά πόσον και η Κομισιό μας έδωσε μια πολύ καλή και ακριβή εικόνα. Θα δούμε κατά πόσον τα τεχνικά στοιχεία και τα νέα τεστ, milestone τεστ θα είναι επιτυχή. Αλλά ε, θα ήταν όλα τα πράγματα καθόλου θετικά. Ωραιότατα. Λοιπόν, ψηφίζουμε αυτή τη μεταφορά υπαριθμών 18 που τη συστήνει ένθερμα εισηγήτρια. Ποιος είναι υπέρ. Μεταφορά 18. Ποιος είναι υπέρ. Ξυπνήστε. Ε. Κατά. Μία αποχές. Η 18 εγκρίνεται. 19 πρόκειται για μεταφορά για ανθρωπιστική βοήθεια προς το μέσο ανθρωπιστικής βοηθείας και για δράσεις στη Λιβύη και στην ακτή του Ελεφαντοστού. Πριν πάρει το λόγο η συγγήτρια να διευκρινίσω ότι στη σελίδα 7 του εγγράφου ο όρος που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, in the northern part of Cyprus, θα πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο, τον πολιτικά ορθό, τον εξή. Σε αυτές τις περιοχές της Δημοκρατίας της Κύπρου, στην οποία η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, πραγματικό έλεγχο. Ο καθένας κατανοεί την απόχρωση ε, και δεν, είναι, δεν αφορά τον προπολογισμό, αλλά η διατύπωση είναι πάρα πολύ σημαντική πολιτικός πώς Όσον αφορά αυτή την πρόταση μεταφοράς, κυρία Συγήτρια, ποια είναι η πρότασή σας. Η σύστασή μου θα ήταν να υπερψηφίσουμε. Δικαιολογείται, σωστό το αίτημα, ξέρουμε ότι ακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις και στην ακτή του ελεφαντοστού και στη Λιβύη και δεν έχω επιφυλάξει ούτε για το ποσό. Άρα είμαι υπέρ. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς υπαριθμών 19. Σας ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα έχουμε άλλη τώρα μια ψηφοφορία που αφορά το, την πρόταση μεταφοράς 5 και 10, Της μεταφορές 5 και 10 αλλά κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματο της Επιτροπής Απασχόλησης που πρέπει να γνωμοδοτήσει και ψηφίζει μόλις το απόγευμα, προτείνω να αναβάλουμε αυτή την ψηφοφορία για το τέλος της σημερινής συνεδριάσεώς μας, για την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για δύο, σε δύο τομείς, έκθεση Ματέρα και Ράιμερ Μπέγκερ, η Επιτροπή Επασχόληση λοιπόν ψηφίζει αρχέ του απογεύματο και από ευγένεια προς την Επιτροπή αυτή θα ψηφίσουμε εμεί το τέλος του απογεύματο. Ευχαριστώ τη Σιδόνια. Έχουμε μία μεταφορά, τουλάχιστον φορά, το προϋπολογισμό των άλλων θεσμικών οργάνων, η Helga Trippel, Helga, η οποία είναι πολύ χαροπή, η μεταφορά αυτή την χαροπή, θα μπορούσε ίσως να μην αρκείτε να μοιράσετε τη χαρά σας με τον Ράιμερ Μπέγκε και να μας παρουσιάσει το θέμα. Χέλγα, Χέλγα, είμαστε τόσο χαρούμενοι που σε βλέπουμε, λέει αγγλιστή ο πρόεδρος, τόσο χαρούμενοι. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα εσύ ως εισηγήτρια να μας παρουσιάσεις σχέδιο της προτάσεις μεταφοράς για τα άλλα θεσμικά όργανα ούτως ώστε να είναι όλοι χαρούμενοι και γελαστοί. Εντάξει, μισό λεπτό. Πρόεδρος, ε, έχουμε πρόταση μεταφοράς για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. C4. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει η κυρία Τρίπελ. Έχουμε δύο τίματα οι μεταφορέ. Ξεκινήσουμε με το λιγότερο προβληματικό θέμα, τη λιγότερο προβληματική μεταφορά, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Πρόταση που επιβλήθη προ εξέτασή μα γενική μεταφορά. 14 γραμμέ του προπολογισμού αφορά. Δεν θα αναφέρουμε κάθε μεταφορά. Ο όγκος συνολικός είναι 5,5 εκατομμύρια ευρώ συνολική μεταφορά. Βασικά γραμμές, βασική μισθή, αμοιβέ και δικαιώματα του μονίμου προσωπικού. Ενισχύσει αφορούν κονδύλια, δικαιώματα σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικού που αφορά τις προσωπικές περιστάσεις που αφορούν το προσωπικό. Ε, διενεμήθη λεπτομερής αιτιολόγηση για τη μεταφορά από την αρμόδιο φορέα και αυτό είναι κάτι που το καλοδέχομαι. Βασικός λόγος που αναφέρεται στον προπολογισμό αυτό πρέπει να προσαρμοστεί ο προπολογισμό, διότι κάποιε γραμμέ του προπολογισμού είτε είχαν υπερεκτιμηθεί είτε υποεκτιμηθεί όταν είχε καταρτιστεί ο προπολογισμό το 2010. Αυτό είναι κατανοητό, διότι είναι δύσκολο να προβλέψει κανεί τις ακριβείς ανάγκες ενός νέου φορέα, ενός θεσμικού οργάνου νέου. Εγώ προτείνω να δώσουμε πράσινο φως σε αυτή την ε, μεταφορά. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ζητά κανείς το λόγο. Πολύ καλά. Λοιπόν, υποβάλλουμε την πρόταση μεταφοράς στη ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς αυτής. Μεταφοράς για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχει αποχή. Οπότε η μεταφορά υπαριθμών 2 2011 για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη μεταφορά C4 που αφορά το κοινοβούλιο μας. Ευχαριστώ λέει κυρία Τρούπελ. Όσον αφορά τη δεύτερη μεταφορά έχω κάποια προβλήματα. Η μεταφορά αφορά το δικό μας ε, οίκο και αφορά περιθέσω το θεματικό 5 εκατομμυρίων ευρώ για εφαρμογές πληροφορικής αποφάσισε πέρσι το Κοινοβούλιο να διαθέσει αυτό το ποσό στο αποθεματικό, αναμένοντας περισσότερες πληροφορίες περί του προγράμματος κινητικότητας πληροφορικής και ζητήσαμε εμβριθέστερη ανάλυση και συζήτηση. Η πρώτη προϋπόθεση πληρείται κατά απόψή μου, αλλά παρακολούθησα και μια γενικότερη συζήτηση που διεξήχθη επί του θέματος. Ε, μάλλον δεν, δεν συμμετείχα σε τη συζήτηση, οι συνάδελφοι να γνωρίζουν έχω κάποια προβλήματα, έχει περάσει ο χρόνος και φαντάζομαι ότι περιμένει η δίκηση τα χρήματα. Αυτό είναι το ένα. Απ' την άλλη είναι και θέμα αρχής όμως, διότι υπάρχει κάποια τάση στη δίκηση να αποφεύγει τις συζητήσεις πέρα από το επίπεδο Προεδρείου για θέματα που πολύ συχνά όμως είναι σημαντικά και αφορούν πάρα πολύ κόσμο και πάνω απ' όλα ε, είναι δαπανηρά. Άρα θα με ενδιέφερε να ξέρω ποιες είναι οι εντυπώσεις των παρόντων συναδέλφων. Προσωπικά μπαίνω στον πειρασμό να αναβάλω αυτή τη μεταφορά ε, λόγω αυτών των συνθήκων. Για να συνοψίσω λοιπόν, ε, βλέπω ότι υπάρχει έλλειψη συζήτησης εδώ, αλλά αυτό για αυτό που θέλουμε και να πω και κάτι άλλο. Στις πληροφορίες που πήραμε μέχρι τώρα υπάρχει μια πρόταση. Να έχουμε την ε, δυνατότητα πληροφορικής στην Ορομέλεια και αλλού, να έχουμε Wi-Fi αλλά γίνονται πολλές βιντεοδιασκέψεις εντός κοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν χρειάζεται αυτό. Διότι πολλοί συνάδελφοι τελικά ίσως να μην έρχονται στις συνεδριάσεις και να κάνουν βιντεοδιασκέψεις εντός του κοινοβουλίου και αυτό δεν είναι καλό για το κοινό, ε, για τον κόσμο. Και θέλω να το συζητήσω κατά πόσο το χρειαζόμαστε αυτό. Ίσως θα ήταν μια καλή λύση να μην πάρουμε όλο το αποθεματικό, αλλά ένα κομμάτι του αποθεματικού, αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ακούσω ποιε είναι οι απόψει των συναδέλφων μου περί αυτού. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Χέλγα. Γκόραν Φέρμ είναι έτοιμο να δώσει μια απάντηση σε αυτά που υπόθηκαν. Μερικά σχόλια. Συμφωνώ με τη Χέλγα, είναι λίγο δύσκολο διότι έχουμε λάβει πολλές πληροφορίες, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε στατηγικά το θέμα, συμφωνώ μαζί της. Υπάρχουν ένα-δύο πράγματα που πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητηθούν. Παραδείγματο χάρη, τι γίνεται με το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη της τονοποιημένου προγράμματος ε, επικοινωνία. Ξέρουμε ελάχιστα μακρόν το επεξεργάζονται, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Τι γίνεται με την άλλη ιδέα για λιγότερο, μικρότερη χρήση χαρτιού στις κοινοβουλευτικές μας συνεδριάσεις. Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες επ' αυτού, τι μπορούμε να πετύχουμε, τι μπορούμε να εξοικονομήσουμε, άρα χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες. Ξέρω ότι έχουμε μέλη στη δική μου ομάδα αλλά και σε άλλες ομάδες που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να δούμε ε, ποιες είναι οι σχέσεις με τη Microsoft. Ε, μήπως πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις στο μέλλον που να βασίζονται σε πιο ανοιχτό κώδικα. Πρέπει να συζητήσουμε κανένα δύο πράγματα πριν το εγκρίνουμε αυτό. Ίσως θα έπρεπε να το θέσουμε σαν σημείο στην ημερήσια διάταξη για μία από τις επόμενες συνεδριάσεις μας. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ο κ. Ενάντες. Η δική μας θέση επί της αρχής είναι υπέρ των στόχων αυτής της μεταφοράς. Νομίζω ότι αυτή τη θέση τη συμμερίζονται και οι υπόλοιπε ομάδε. Είναι σαφές ότι τα ε, συνεχή και περιτά ταξίδια ε, δημιουργούν ε, πρόσθετες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, οπότε μάλλον θα πρέπει να είμαστε υπέρ των βίντεο συνεδριάσεων. Ε, δεν θέλουμε λοιπόν να εκφραστούμε εναντίον του, του project αυτού, ας εμβαθυνθεί η συζήτηση. Παρ' όλα αυτά οι πληροφορίες που μας έχουν δοθεί πιστεύω ότι είναι επαρκής, επαρκώς σαφείς και νομίζω ότι ε, δικαιολογούν τη λύση μιας αποφάσεως. Παρ' όλα αυτά, παρόλα αυτά λέω, δεν είμαστε αντίθετοι με την περαιτέρω και σε περισσότερο βάθος συζήτηση του ζητήματος αυτή η αναβολή, υπό την προπόθεση ότι αυτή η αναβολή δεν συνιστά αμφισβήτηση του στόχου. Ευχαριστώ. Très bien. Donc, euh, Λοιπόν, Χέλκα, δεδομένων όσων είπατε εσείς και αυτών που είπαν και οι συνάδελφοι, κατανοώ ότι προτιμάτε να αναβληθεί η ψηφοφορία και ότι μέχρι τότε θα θέλετε οι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου να σας δώσουν διευκρινήσει πάνω στο σημείο που ακόμα δεν είναι απόλυτα σαφή. Λοιπόν, ο πολιτικός στόχος δεν αμφισβητείται, το υπενθύμησε δικαίως ο κ. Φενάντες. Χρειαζόμαστε όμως περαιτέρω διευκρινήσεις. Προτείνω λοιπόν να αναβληθεί η ψηφοφορία για την ε, μεταφορά αυτή. Θαυμάσια. Τώρα, ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες υπό την επιφύλαξη της τελευταίας ψηφοφορίας για την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η Μόνικα δεν έχει έκθεση σήμερα. Θα έχει άλλες ευκαιρίες βέβαια να μας παρουσιάσει την έκθεσή της και μπορούμε να περάσουμε στην εξέταση των δύο εκθέσεων του Καλχαλούντ για τα σημεία 8 και 9. για το πρόγραμμα πλαίσια έρευνα. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για μια ανταλλαγή απόψη. Ίσως θα μπορέσετε να μας παρουσιάσετε και τις δύο εκθέσεις ταυτόχρονα. Για να έχουμε μια κοινή συζήτηση και στα δύο θέματα. Κύριε Χαγκλούτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την οξύ μου στην τελευταία συνέντευξη που συζητήθηκε για το θέμα, γιατί ήμουν αναγκασμένο να πάω στην πατρίδα μου και ευχαριστώ τη συνάδελφο κυρία Γένσεν που με αντικαθέστησε. Η πράσινη βίβλο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα θέμα πολύ ευθυγραμμισμένο με αυτό που συζητήσαμε πλειστάκι στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας τα περασμένα χρόνια. Το σχέδιο γνωμοδότηση που παρουσιάστηκε την περασμένη φορά έχει ορισμένα κύρια θέματα που θέλω να θίξω. Καταρχήν, ότι εκτό από την ιδέα να συνδεθεί η στρατηγική του 2020 με όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα διευθυντικά ταμεία και τομεία συνοχή συνοχής είναι συμπληρωματικά με τη γραμματοδότηση της έρευνας και γι' αυτό δεν χρειάζεται να υπάρχει κάτι το ξεχωριστό. είναι σημαντικό να το τονίζουμε αυτό, νομίζω. Επίση, προσπάθησα στην γνωμοδότησή μου να αναφερθώ στα καινοτομικά χρηματοδοτικά ε, μέσα που εισήγαγε η Κομισιόν, να τα παρουσιάσω θετικά. Υπάρχει κάτι που δεν είμαι πολύ πεπισμένο, ήταν λεγόμενα soft loans, είμαι κάπως επιφυλακτικός Ξέρω ότι ο σκιώδης ηγητή στην σοσιαλιστική ομάδα είναι πιο θετικό και εγώ είχα ζητήσει από την Κομισιόν και την IAB, την Τράπεζα Αναπτύξεως, να μου δώσει περισσότερες εξηγήσει. Και θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε την γνωμοδότηση βάσει τροπολογιών κατόπιν συζητήσεων με την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως. Επίσης θα ήθελα να υπάρχει ένα σύστημα προσέγγισης που βασίζεται στην ε, εμπιστοσύνη, μεγαλύτερη ανοχή δηλαδή κινδύνου. Υπάρχει επίσης το θέμα που έχει θίξει η κυρία Γκρέσλε, θέματα του δημοσιονομικού κανονισμού. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό για να είμαστε επιτυχείς με το 8ο ε, πρόγραμμα πλαίσιο. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που με κάνει να περάσω στη δεύτερη μου έκθεση είναι το θέμα των μεγαλύτερων προγραμμάτων όπως το Ήτριο και το Γαλιλαίο. για να αποφύγουμε τον κανιβαλισμό επί του εβδόμου προγράμματος πλαισίου. θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση που θα μας κάνει να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση. Και τέλος, αλλά πάρα πολύ σημαντικό θέμα, τονίζουμε το γεγονός ότι γενικά χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για την ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής αν θέλουμε να είμαστε πολιτικοί. Αυτό είναι κάτι που τη χάνει πολιτική υποστήριξη. Και ξέρουμε ότι στην ψήφο που δώσαμε στο Στρασβούργο την περασμένη φορά για την έκθεση του κ. Γκαρίγκα ακολουθούμε ακριβώς αυτή τη γραμμή. Αυτό λοιπόν είναι ευθυγραμμισμένα με την έκθεση που πέρασε στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα. Αυτά στα σύντομα για την γραμμοδότηση αυτή. Για την άλλη, επί της στα ε, αρμόδια επιτροπή δεν έχει ακόμα δώσει ε, ένα χρονοδιάγραμμα. Εξαρτάται από την Ήτρε Είμαστε λοιπόν εδώ ευθυγραμμισμένοι, αλλά δεν υπάρχει ακόμα σχέδιο γνωμοδότησης. Δεν θα είναι μακρά βέβαια, αυτό που μπορούμε να προβλέψουμε ήδη είναι ότι υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί το ποσό 100 εκατομμυρίων ευρώ γιατί και οι Ιάπωνες θα μειώσουν τη δική τους χρηματοδότηση και όλοι οι άλλοι θα κάνουν το ίδιο λόγω των, ε, της καταστροφής από το τσουνάμι στην περιοχή του Φουκουσίμα. Θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική υποστήριξη και ότι χρειάζεται να μεταφέρουμε τα κονδύλια στο τομέα της πυρηνική ασφάλειας, κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ το σώμα και αυτό θα πρέπει να το πούμε λοιπόν όταν τελικά υπάρχει ένα ε, κείμενο για δεύτερη αυτή γνωμοδότηση για τη Eurotom. Σε δύο λόγια αυτά κύριε Πρόεδρε για τις δύο γνωμοδοτήσεις. Για την πρώτη έχουμε αρκετά προχωρήσει. Η προθεσμία υποβολή ε, τροπολογιών αύριο, 16 Ιουνίου, και θα εξακολουθώ να συνεργάζομαι με τι άλλε ομάδε για να ολοκληρώσω τη γνωμοδότηση αυτή. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, και σα ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Πάρα πολύ σαφή η παρουσίασή σα. Υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια από συναδέλφους πάνω στην παρουσίαση αυτή. Ο Ράιμερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλω να εκφέρω μια γνώμη γλίγορα σε αυτό που είπε και ο Καλ για την Ήτα και τα προβλήματα που έχουν μείνει άλυτα όσον αφορά την χρηματοδότηση. Δεν ξέρω πώς είτε η Κομισιόν είτε και οποιοδήποτε άλλο θα μπορέσει να ε, αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Θα αρχίσω μια περίγεια εμπειρία που είχα την περασμένη εβδομάδα. Την πέμπτη το πρωί πήρα ένα email από μια γενική διεύθυνση που ασχολείται με το θέμα αυτό, αυτούς που είναι αρμόδιοι για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο μεταξύ 9 και 10 την πέμπτη το πρωί παρακαλώντας ότι ένα σημαντικός ε, ε γενικής διευθυντής, όχι του προπολογισμού, αλλά κάποιος άλλος θέλει να συζητήσει μαζί μου την Πέμπτη το απόγευμα ή την Παρασκευή το πρωί, γιατί την επόμενη εβδομάδα πρέπει να πάει στο Συμβούλιο Ήτερ στην Ιαπωνία. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, πόσο ηλίθιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Πόσο ηλίθιοι είναι. Πώς νομίζουν ότι μπορούν να συμπεριφερθούν έναντι ενός βουλευτή. Εντάξει. Να καταλάβει κανένας ότι πριν από διεθνείς διασκέψεις θα πρέπει να έχουν μια έντονη επαφή με το Κοινοβούλιο και ιδίω με τις αρχές της υπεύθυνης για τον προορισμό πριν να αναλάβουν κάποιες διεθνείς ε, ε, υποχρεώσεις όπως η τέος επίτροπο επίτροπος ε, κυρία Βάλτνερ Φεραίρο Βάλτνερ το έκανε πριν από τη συμμετοχή της στις ε, διασκέψεις των δωρητών. Ωραία. Αλλά όχι έτσι. Δεν είναι τρόπος αυτός να μας αντιμετωπίζουν. Ε. Ταυτόχρονα δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχουν δυνατότητες το Συμβούλιο πριν από τις διακοπές να συμφωνήσει πάνω σε μια λογική πρόταση πώς σκοπεύουν να χρηματοδοτήσουν την ΙΤΕΡ. Το σχέδιο αυτό ΙΤΕΡ. Συζητιέται αναθεώρηση, μεταφορά, συμπληρωματική χρηματοδότηση. Εγώ άκουσα ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που διαφυσβητήσουν όλο το ποσό. Λένε μήπως θα έπρεπε να είναι κάπως λίγο, λιγότερο. Άλλοι λένε «Α, όχι, για να περιμένουμε να ολοκληρωθεί στις 15 Οκτωβρίου το ε, οικονομικό έτος της Γεωργίας για να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχουμε και τώρα και την για τα οπορικαιοφυτικά και δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα που δεν θα έχουν δαπανηθεί. Και όλα αυτά θα πρέπει να προσαρμοστούν ούτως ώστε ο προβλησμός 2012 να έχει τη μορφή που θέλουμε. Την τρέχουσα εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά ποιες είναι οι συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό και εν ώψη του τριμερούς διαλόγου του Ιουλίου. Γιατί αυτό που δεν επιτρέπει να συμβεί είναι η ανικανότητα του Συμβουλίου να υπάρξει ξεχωριστή απόφαση για το σχέδιο ΙΤΕΡ να οδηγήσει σε συνένωση διαφόρων θεμάτων που θα έχουν τελείως ανωτικό αποτέλεσμα και μετά να η εντύπωση ήταν είναι υπεύθυνο το κοινοβούλιο για αυτά. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά την ομοφωνία στις ε, ε αναθεωρήσεις του προβολισμού τι γίνεται. Δηλαδή, αυτές οι τροποποίησεις που θέλει να επιβάλλει το Συμβούλιο λόγω της δήλωσης στα πρακτικά της συνθήκης της Λισαβόνας, θα πλήξει τελικά το Συμβούλιο το ίδιο, γιατί εμείς δεν θα συμφωνήσουμε πάνω στην διαδικασία, στην συνθήκη της, συγγνώμη, στη διαδικασία βάσης της συνθήκης Λισαβόνας. Και ίσως πριν από τον τριμερή διάλογο θα ήταν καλό να ασχοληθούμε με το θέμα, ίσως και κεκλεισμένο των θυρών και μετά ίσως θα πρέπει να αποταθούμε προς την κοινή γνώμη μετά από ε, εις βάθος συζήτηση με τους ε, συντονιστές ούτως ώστε τελικά η αδυναμία δράσης του Συμβουλίου και η αρνητική στάση της Κομισιόν να μην οδηγήσει το να είμαστε εμείς τελικά οι θεωρούμενοι υπεύθυνοι για την αποτυχία. Και σας το λέω αυτό εν ώψη αυτά που βλέπουμε να γίνονται ε, στο Συμβούλιο και από την Κομισιόν επίσης που κατά τη γνώμη μου το Συμβούλιο δεν εργάστηκε πολύ σοβαρά με τα αριθμικά στοιχεία που έχει στα χέρια του. Ευχαριστώ, Ράιμερ. Η Αν Γέντσεν έχει το λόγο. Well, I'd like to thank for... Ευχαριστώ τον Ράινερ για αυτές τις ε, διευκρινήσεις. Παρόλο που η κατάσταση δεν είναι και πολύ σαφής. Ως ε, συνεπικεφαλής της αντιπροσωπείας που στείλαμε να, δουν, να δούμε τον Ίτερ, ε, ε, πήρα μια επιστολή από τον Επιτροπό Κουίν που μας ε, πιέζει. Η Κομισιόν γενικότερα μας πιέζει. Συνεπώς θα χειροκροτούσα, συμφωνώ δηλαδή με την πρόταση του Ράινερ να το δούμε σε, λίγο ε, έτσι ώστε η απάντηση να προέρθει από τον πρόεδρο τον ίδιο. Στο Κανταράς το είχαμε συζητήσει και από τότε είχαν φανεί οι δυσκολίες γιατί το πρόβλημα από πλευράς του Κοινοβουλίου δεν είναι απαραίτητα το ίδιο το project αν εξαιρέσουμε τους πράσινους αλλά η χρηματοδότησή του το γεγονός δηλαδή ότι η Κομισιόν πρότεινε ένα μεγάλο τμήμα της χρηματοδότησης να προέλθει από, ε, ερευνητικά, από τον προπολογισμό ερευνητικών προγραμμάτων. Τώρα βέβαια, το Συμβούλιο έχει αλλάξει στάση, ήθελε στην αρχή όλος ο προπολογισμό να προκύψει από τον ε, από τα ερευνητικά σχέδια, αλλά ακόμα και έτσι είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε εμεί εδώ από πλευρά Κοινοβουλίου. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να ε, πάρουμε μια εύκολη γρήγορη απόφαση. Ε, από την άλλη μεριά έχουμε και το Συμβούλιο το οποίο αργεί. Ίσως η Κομισιόν θα έπρεπε να πιέσει και το Συμβούλιο να, να λογικευτεί λιγάκι και όχι μόνο να πιέζει εμάς συνεχώς. Ευχαριστώ, κύριε Καρβάλιο. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή να εστιαστώ στο κοινό, στο τμήμα που αφορά το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Συμφωνώ με την έκθεση του εισηγητή που μας την παρουσίασε κιόλας. Ε, επιπλέον, των σχολείων του εισηγητή. Όμω θέλω να υπογραμμίσω και το εξή. Την σημασία του να δημιουργήσουμε ένα οδικό χάρτη για τον στόχο του 3% για τις επενδύσεις σε project ε, έρευνας και καινοτομίας. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε καλή διακυβέρνηση τόσο σε επίπεδο της Κομισιόν όσο και επίπεδο κρατών μελών στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Η αυτή είχε, έχει προστεθεί, έχει συμπεριληφθεί και στην έκθεση ΣΟΥΡΕ, οπότε καλό θα ήταν να το τονίσουμε και εδώ, το πόσο σημαντικό δηλαδή είναι το 3% και το πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτό το 3% σε επενδύσεις ε, έρευνας και καινοτομίας. Και κάτι άλλο σχετικό, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο ε, εστιάζεται στην αριστεία και ε, συμπληρώνει τα διαρθρωτικά, τις διαρθρωτικές δράσεις, τα διαρθρωτικά ταμεία. Χρειάζεται να εξασφαλιστεί αυτή η συμπληρωματικότητα και ε, συμβατότητα των κανόνων τους. Ε, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζονται πολύ διαφορετικούς κανόνες υπάρχουν χώρες στις οποίες οι ερευνητές έχουν πρόσβαση στα ερωτικά ταμεία και ε, κάνουν αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση από το στρατηγικό πλαίσιο, αλλά έχουν τόσο πολύ διαφορετικούς κανόνες που δυσκολεύονται. Μια και απλοποιούμε το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και τους κανόνες του, θα έπρεπε να δούμε και την απλοποίηση της χρηματοδότησης που προέρχεται από τα διαφορετικά ταμεία. Ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν μέσα τα οποία είναι γρήγορα, ελαστικά, εύκολα να χρησιμοποιηθούν στο κοινό πρόγραμμα. Το κοινό πρόγραμμα μέχρι σήμερα είναι πολύ περίπλοκο. Συνεπώς, θέλουμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να αναζητήσει αυτούς τους ευκολότερους, πιο ελαστικούς τρόπους ε, για να ε, κάνουμε πιο ρέουσα τη σχέση ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο. Αυτά επιπλέον των όσων είπε ο Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. James Ellis. Ε, ευχαριστώ τον εισηγητή και για τα δύο αυτά θέματα. Είναι εξαιρετικά ε, σημαντικό αυτό το ζήτημα για τη μελλοντική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ε, το θέμα του κινδύνου και της απλοποίησης ε, επανέρχεται συνεχώς. Ε, θα πρέπει να ξανακερδίσουμε αυτούς τους ερευνητές οι οποίοι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία εξαιτίας της πολυπλοκότητας των κανόνων. Ας αποφύγουμε λοιπόν την απώλειά τους. Ε, δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ίτερ, έχω δύο σχόλια. Καλωσορίζω τα αποτελέσματα της επίσκεψης. Δυστυχώς εγώ δεν κατάφερα να είμαι μαζί σας, διάβασα όμως την έκθεση η προσέγγιση της ε, αποστολής μας ήταν πάρα πολύ λογική, αν εξαιρέσουμε τα δύο άκρα, ε, πολύ λογική και ιδιαίτερα για τη χρήση των κονδυλίων. Ε, με ανησυχεί όμως τα όσα είπα ο Ράινερ για την διαδικασία που θα ακολουθεί σε επόμενες εβδομάδες. Αν κατάλαβα καλά, υπάρχει ένα project, το JET, ε, στην δική μου εκλογική περιοχή, η περιφέρεια, ε, το οποίο σταδιακά θα καταργηθεί ίσως μέχρι το 2014-2015. Εκεί όμως έχουμε μαζεμένους ε, πάρα πολλούς εμπειρογνώμονες με πολύ εμπειρογνωμοσύνη, οι οποίοι θα έπρεπε να βοηθήσουν το στήσιμο του ΙΤΕΡ. Σιγά σιγά φοβάμαι ότι θα τους χάσουμε όμως, διότι το ΙΤΕΡ ε, μάλλον η απόφαση για το ITER δεν έχει ληφθεί και δεν πρόκειται να ληφθεί ενδεχομένω ούτε μέχρι το 2012. Εν τω μεταξύ, το JET χάνει τα, τον προπολογισμό του, μειώνεται ο προπολογισμό του, οπότε φοβάμαι θα χάσουμε του επιστήμονε αυτού. Συνεπώ, ε, όταν φτάσουμε στον τριμερή διάλογο, μέχρι να φτάσουμε στον τριμερή διάλογο, α συμφωνήσουμε ε, για τον προπολογισμό του 2012 για αυτό το ζήτημα. Έχουμε δύο χρόνια μετά μέχρι την, ε, ε, το κλείσιμο του JET ε, αλλά ας καταφέρουμε μέχρι το 2012 να συμφωνήσουμε πριν το καλοκαίρι γιατί φοβάμαι ότι το φθινόπωρο θα, αρχίσουν, θα αρχίσει το προσωπικό να διαρρέει από το JET και θα το χάσουμε. Ευχαριστώ James. Το διακύβωμα είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Το είπανε πολύ ιδιαίτερα ο Ράινερ. Είναι ανησυχητική εξέλιξη του θέματος ίτερ. Ε, και εγώ ίδιος ανησυχώ πολύ και με ανησυχεί το γεγονός ιδιαίτερα ότι το Συμβούλιο δεν ξέρει τι θέλει. Έχοντας, ε, λαμβάνοντας υπόψη τελευταίες εξελίξεις, στο επιστημονικό αλλά και το δημοσιονομικό και το πολιτικό επίπεδο, το Συμβούλιο φαίνεται να μην ξέρει πια τι θέλει. Οπότε, έσαφες ότι αν η χρηματοδότηση των νέων δαπανών, του πρόσθετου κόστους δηλαδή του ΙΤΕΡ, θα πρέπει να προέλθει α, μόνο από το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, τότε το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα θα απολέσει την κρίσιμη μάζα που είναι απαραίτητη για να είναι χρήσιμο σε άλλους τομείς. Δηλαδή θα θυσιάσουμε τα πάντα στο βωμό του Είναι χρήσιμο το Twitter, ασφαλώς, αλλά δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει, να προοδεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η αποτελεσματικότητά της, η καινοτομία της, η Ατζέντα Ευρώπη 2020 και όλα αυτά ε, με ε, μια μειωμένη χρηματοδότηση και με χρηματοδότηση, πλήρη χρηματοδότηση μόνο των μεγάλων project. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα εκεί. Αν έχω καταλάβει καλά, η Ουγγρική Προεδρία και η Πολωνική Προεδρία κατόπιν θα υποβάλουν καινούργιε προτάσεις στο Συμβούλιο, στο αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών. Συνεπώς στι επόμενες εβδομάδες και στι επόμενε μέρες θα δούμε εξέλιξει. Και όπως είπε ο ε, Ράιμερ, Ε, θα πρέπει να συζητήσουμε τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε έτσι ώστε να δούμε πώς το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας μπορούν να λάβουν θέση ε, από τακτικής και πριν τον τριμερή διάλογο γιατί χτες το βράδυ το συζητήσαμε με τους συντονιστές. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι πως το θέμα αυτό θα έρθει στην ημερήσια διάταξη του τριμερούς διαλόγου είτε το προτείνει το Κοινοβούλιο είτε όχι γιατί είναι ένα θέμα της επικαιρότητα. οπότε θα πρέπει να έχουμε θέση μέχρι τότε, θα πρέπει, να, θα πρέπει να έχουμε τοποθετηθεί μέχρι τότε. Μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα γίνει την επόμενη Δευτέρα. Στο πλαίσιο της ε, κοινή ε, συνεδρίασης Επιτροπής ΣΟΥΡΕ και της δική μας Επιτροπής, ε, παρουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής και κλεισμένων των θυρών, το λέω αυτό σε όσους συμμετέχουν σε εργασίε μας χωρίς να είναι μέλη της Επιτροπής Προπολογισμών, θα είναι και κλεισμένο το θερών αυτή η συνεδρίαση της επόμενης Δευτέρας. Κοινή συνεδρίαση μεταξύ των ε, βουλευτών που ασχολούνται με το ζήτημα στην Επιτροπή Προπολογισμού, προσκαλώντας και την Επιτροπή ΣΟΥΡΕ. Τη Δευτέρα θα δούμε ε, πού βρίσκεται το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ταυτόχρονα ε, θα εξετάσουμε και αυτό το ζήτημα Twitter. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Ο κύριος, ε, κύριε Χάγκλοντ, θα βγάλουμε συμπεράσματα από αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά καταρχήν τη, την πράσινη βίβλο του νέου πρόγραμματος πλαισίου, θα συμφωνήσω με την κυρία Καρβάλιο. Ε, μέχρι αύριο ε, θα έχουμε έτοιμες τροπολογίες. Ιδιαίτερα το θέμα του οδικού χάρτη θα το λάβουμε υπόψη διότι υπάρχει, εξασφαλίζει συνένεση. Μετά, για το θέμα του Twitter. Συμφωνούμε με τους συναδέλφους Μπέργκ και Γέντσεν. Συμφωνώ. Καθώς επίσης και με τα συμπεράσματα τα δικά σας, Πρόεδρε. Στον James ε, Ellis να πω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να βρεθούμε κατηγορούμε ότι είναι δική μας ε, ευθύνη η, η μείωση της χρηματοδότηση. Γιατί το Συμβούλιο και οι Κομισιόν δεν έχουν δράσει ικανοποιητικά μέχρι τώρα και τώρα αυτό που μας ζητούν είναι να μειώσουμε τον προπολογισμό των άλλων προγραμμάτων έρευνας. Θα πρέπει να αποφύγουμε επίσης να βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση στις εκλογικές μας περιφέρειες. Ε, Ας ε, ε, μην γίνουμε από δύο πομπέι τράγοι. Καλό είναι λοιπόν να γίνει μια στρατηγική συζήτηση για το πώς θα χειριστούμε το θέμα και κλεισμένο των θυρών ε, στην ε, περίπτωση που δεν θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Πιστεύω ότι είναι αδύνατο να πάρουμε από το πρόγραμμα πλαίσιο τη έρευνα τόσα ποσά όσα ζητάει το Συμβούλιο. σω μπορέσουμε να βρούμε βέβαια μια διάμεση λύση. Πάση περιπτώσει όμω η πρόταση που έχουμε αυτή στην μπροστά μα δεν είναι αποδεκτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί βάση για συμφωνία. Αυτό νομίζω το πιστεύει ε, η μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Ευχαριστώ. Merci, Πολύ καλά. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Να ότι όσον αφορά την πράσινη βίβλου για το στατικικό πλαίσιο της έρευνας. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 16 Ιουνίου στις 1 το μεσημέρι και θα πρέπει να εθετήσουμε την έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στη συνεδρίαση της 12ης και 13ης Ιουλίου εν ώψη προετοιμασίας ψηφοφορίας που θα λάβει η χώρα στην ΕΤΡΕ στις 30 Αυγούστου και στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου, τη δεύτερη σύνοδο του Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά την άλλη έκθεση για τα πυρηνικά, υποθεσμία, για τις τροπολογίες ήδη πέρασε και η ψηφοφορία θα πρέπει να γίνει στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Ωραία, αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούν πιο γρήγορα, αυτό το καλύτερο, κερδίζουμε και χρόνο. Σας προτείνω λοιπόν να πάμε στο σημείο 12. Ε, ο συνάδελφος Κοτσολίνο είναι εδώ. Λοιπόν, σας δώσω το λόγο. Για τα άλλα μέλη της Επιτροπής Περιπολογισμού να πω ότι δουλέψαμε τόσο καλά που έχουμε αρκετά σημαντική επιτάχυση των εργασιών. Λοιπόν, τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως της Σερβίας θα τον προειδοποιήσω ότι είμαστε έτοιμοι για την ακρόαση στο πρώτο τμήμα της απογευματινής συνεδριάσεως. Προτείνω να προχωρήσουμε τώρα στην έκθεση Κοτσολή, να προσπαθήσουμε κατά τις 10.30 να έρθει ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως ο Σέρβος και στις 15.30 και θα ψηφίσουμε την έκθεση Μπάρμπαρα αμέσως μετά. Θα εξηγήσουμε στην Επιτροπή Απασχόλησης ότι ψηφίσαμε... Πότε ψηφίσαμε, τέλος Λοιπόν, έτσι θα το ολοκληρώσουμε πιο νωρί τι εργασίε μα. Νομίζω ότι είναι προ συμφέρον όλων. Βέβαια, έχουμε την έκθεση του κυρίου Σουριάν και θα δούμε αν μπορέσουμε ήδη να την εξετάσουμε το πρωί ή αρχέ του απογεύματο. Πρώτα απ' όλα ο κύριο ε, Κοτσολίνο και μετά ο Λάσλο. Και ανάλογα με το χρόνο που θα χρειαστούμε για τον κύριο Κοτσολίνο, ο Λάσλο θα μπορούσε να παρουσιάσει την έκθεσή του το πρωί ή αρχέ του απογεύματο. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Συμφωνείτε, ευχαριστώ. Κύριε Κοτσολίνο, λοιπόν, Έχετε το λόγο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πάρα πολύ σύντομα. Πρέπει να εκφράσουμε μια γνώμη επί της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την καταπολέμηση της φτώχειας. Γνωρίζουμε ότι είναι μια από τις προτεραιότητες στρατηγικής για το 2020 και γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε αυτή την πλατφόρμα, δηλαδή ένα πλαίσιο εργαλείων, ένα, μια εργαλειοθήκη για να καταπολεμήσουμε την κοινωνικό αποκλεισμό και την αυξανόμενη φτώχεια στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε επίσης από το πόσο είναι σημαντικός ο ρόλος των κρατών μελών, από αυτά που είπα. Και επί οποίων σημείων πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο την προσοχή μα για να γνωμοδοτήσουμε σε Επιτροπή Προπολογισμών. Θα ήθελα να εστιασώ αυτά που θα πω επί δύο απαιτήσεων. Πρώτον, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνοχή όσον αφορά τι γενικέ δηλώσει που κάνουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν Κοινοβούλιο, σαν κράτη-μέλη με, τα, με τους πόρους που διαθέτουμε ε, όσον αφορά την πολιτική αντίθεσης ε, καταπολέμησης στόχης και του ελληνικού αποκλεισμού. Οι ίδιες συστάσεις που αναγνωρίστηκαν στις 7 Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα πρώτα προγράμματα μεταρρυθμιστικά για τα διαφορα κάτι κράτη-μέλη ε, δείχνει πόσο χρειάζεται τα κράτη-μέλη να, έχουν, να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή και να έχουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα όσον αφορά την δήλωση των πολιτικών που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη για να αντιταχθούν στην φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτές τις μέρες είχαμε διάφορες μεστικές δηλώσεις των διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων που ζητούν από το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να έχουν μεγαλύτερη συνοχή και να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει πάνω απ' όλα να το δούμε αυτό το θέμα σαν Επιτροπή Προπολογισμών επισημάνουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή, μεγαλύτερη σχέση μεταξύ των πολιτικών που ανακοινώνουμε, των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουμε και εν ώψη της στρατηγικής για το 2020 και των συγκεκριμένων πόρων που διαθέτουμε για αυτή την πολιτική. Εν αυτή τη ενία, πέρα από μια έκκληση προς τα κράτη-μέλη, πρέπει να κάνουμε μια έκκληση προς τους ίδιους μας τους εαυτούς. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διότι είναι ασαφές πώς καθορίζουμε το πλαίσιο της Επιτροπής του, το, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ε, τις προτεραιότητες και τη στρατηγική που θα αφιερώσουμε την κατευθύνση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε να αναφέρουμε διάφορα εργαλεία και το 2012 να ζητήσουμε αύξηση του ποσοστού των ποσών που διαθέτουμε για αυτά τα προγράμματα και θα πρέπει διαφανώ να δείξουμε που βρίσκονται αυτοί. Όταν θέλουμε να δώσουμε διαφάνεια στη διάθεση των πόρων, εκείνη είναι δύσκολη δουλειά. Για εμά, την Επιτροπή των Προπολογισμών, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε την πρώτη μεγάλη επιλογή. Να θέσουμε ξεκάθαρα, πιο διαφανώ, πιο ξεκάθαρα το όλο ζήτημα εδώ στο δικό μας επίπεδο, σε επίπεδο κρατών μελών. Και εμείς πώς προσεγγίζουμε την χρήση των πόρων του κοινοτικού προϋπολογισμού για αυτούς τους στόχους. Ε, λοιπόν, δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω στην Επιτροπή είναι εξή. Δεν έχουμε έλλειψη πολιτικών αυτά τα χρόνια. Αυτά τα χρόνια τα ιδιωτικά ταμεία κυρίως ήταν μια πολιτική που καταπολέμησε τη φτώχεια και το κοινωνικό ταμείο και το ταμείο για τους πρόσφυγες και το ταμείο για, τις, για την περιφερειακή ανάπτυξη και όσον αφορά και τι διάφορε συνολικές πολιτικές που εφάρμοσε η Ευρώπη σε αυτούς τους τομεί. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μία επαλήθευση, αν θέλετε. Μία ανάλυση λεπτομερή ε, του ποια είναι η κατάσταση. Γίνονται αυτές οι πολιτικές σε διάφορα επίπεδα. Και έχει δεσμευτεί η Ευρώπη για αυτά, μέσω διαφόρων μέσων που χρησιμοποιεί. Η πολιτική συνοχή χρησιμοποιήθηκε Φερρυπίν και δεν ξέρουμε ακριβώ ποιε συνέπειε έχουν παραχθεί και παράγουν αυτά τα προγράμματα, διότι είναι προγράμματα που είναι καθοδόν, 2007-2013. Λοιπόν, το άλλο σημείο επί το οποίο θα ζητούσα από την Επιτροπή να τοποθετηθεί είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, να γίνει μια εξακρίβωση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του ΣΥΠΗΝ των πολιτικών που μέχρι τώρα ε, δρομολογούμε, χρησιμοποιούμε. Ε, και χρησιμοποιούμε πόρους κυρίως για την πολιτική συνοχή. Εγώ θα συγκέντρωνα, αν θέλετε, διότι είναι γνωμοδότηση που θα πρέπει να ετοιμάσουμε εμείς, σαν Επιτροπή Προπολογισμών, εγώ θα εστιαζόμουν επί των δύο αυτών σημείων. Εκεί θα επικέντρωνα την προσοχή της πρωτοβουλίας μας, της γνωμοδοτήσεώς μας ως Επιτροπή Προπολογισμών, ως συνεισφορά στη μάχη κατά της φτώχειας, κατά, για τη μείωση των κινδύνων του κοινωνικού αποκλεισμού, να κάνουμε πιο διαφανή, πιο ορατή και πιο συγκεκριμένη αυτή τη μάχη για την καταπολέμηση των φαινομένων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Ο κ. Κοσλόφσκι έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ με τον εισηγητή. Είναι πάρα πολύ σημαντική η θέση της Επιτροπής Προπολογισμών να ζητήσει λεπτομέρειες από την Κομισιόν σε σχέση με τη χρήση των ε, πόρων για την πρωτοβουλία αυτή την οποία συζητάμε. Ταυτόχρονα θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτή η πλατφόρμα είναι πολιτής. Άρα χρειαζόμαστε λεπτομέρειες όχι μόνο για το προπολισμό του 2012 αλλά και για τους άλλους δεν μπορούμε να υπερτιμήσουμε ποτέ την σημασία του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και γι' αυτό θα έλεγα ότι αυτή η πρωτοβουλία ε, θα πρέπει να έχει την κύρια σημασία και ο συντονισμός των διαφόρων ταμείων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ταυτόχρονα υπάρχουν και συμπραγματικά στοιχεία. Όταν παραδείγματο χάρη το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Progress που αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου και την ε, δημιουργία και συγκεκριμένη έκφραση ανεφόρων στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην πλατφόρμα. Θα ήταν καλό να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και το ευρωπαϊκό εξάμεινο εδώ, μέσα στα πλαίσια των ελόγων στόχων, λαμβάνοντας υπόψη ότι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας δεν αναφέρονται στην πρόταση της Κομισιόν. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα 75% των δέσεων απασχόλησης δημιουργούνται από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη. Και, η... για να βοηθήσουμε τις απειλόμενες ε, ομάδες θα πρέπει να δούμε ποια σημασία αποκτούν οι νεολαία, οι ηλικιωμένοι σε αυτό το θέμα. Θα ήταν καλό λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μα. Εμεί ε, είπαν οι συνάδελφοι ότι οι μεγάλε πόλει έχουν προβλήματα φτώχεια. Ναι, φυσικά είναι σωστό αυτό. Αλλά ε, θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν παρόμοια προβλήματα και για τους κατοίκους της υπαίθρου που έχουν πολύ δύσκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες και τη δυνατότητα εξέβρεσης θέσεων απασχόλησης. Και από αυτό συχνά υποφέρει και η οικογένεια, τα παιδιά όταν οι γονείς τους είναι ε, άνεργοι ή υπάρχει φτώχεια στην οικογένεια. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Υπάρχει επίσης το πρόβλημα της πρόσφυσης πληροφορίας γιατί δεν υπάρχει το δυνατότητα διαδικτύου. Επίσης θα ήθελα να πω ότι η ένδια είναι πολύ πιο έντονη και μεταξύ των τομέων του πληθυσμού που έχουν ειδικέ ανάγκες. Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω τα μέτρα για την υποστήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της απασχόλησης για τους νέους, τις γυναίκες και τους μετανάστες. Εδώ θα πρέπει νομίζω να υπάρχουν μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης ή μετακπαίδευση που καλύπτουν ακριβώς αυτές τις ομάδες του πληθυσμού που έχουν τα ιδιαίτερα προβλήματα. Γιατί τα προγράμματα παιδείας, μετακπέδευσης κατάρτισης μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν κατά πολέμηση της ανεργίας. Και τελευταίο σημείο. Ε, κατανοώ τις προθέσεις του κ. Σταντέλη, δεν μπορώ να συμφωνήσω πλήρως όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση όλων των εργαζομένων σε όλα τα κρατημέλη. Και δεύτερον, συμφωνώ ότι εκπρόσωποι των ομάδων που πλήττονται από την ένδια χρειάζονται επίσης μια πλατφόρμα ετήσια και υπό Πολωνική Προεδρία στις 17 και 18 Οκτωβρίου θα λάβει χώρα στην Κρακοβία με τέτοια πλατφόρμα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφε, αυτά τα θέματα πολιτικά είναι πάρα πολύ δύσκολα για μας. Γιατί έχουν τεράστια πολιτική σημασία στην εθνική ζωή κάθε χώρα. Πολλές από τις κοινωνικές δυσκολίες που έχουμε στις χώρες μας ε, σχετίζονται με την οικονομική κρίση και για την οικογενειακή κρίση έχουμε προγράμματα τράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καλή λειτουργία τη εταιρεία αγορά, συντονισμό των οικονομικών των κρατών μελών κλπ. Αλλά για την κοινωνική πολιτική έχουμε πολύ λιγότερες νομικές αρμοδιότητες και λιγότερα δημοσιονομικά μέσα. Βρισκόμαστε λοιπόν συνεχώς ενώπιον ενός διλήμματος, όπως το είδαμε στις κύριες ανησυχίες μας, οι πολίτες περιμένουν από εμά να συζητήσουμε κοινωνικά προβλήματα, κρίση, απασχόληση, ένδια, αποκλεισμό. Από την άλλη μεριά, αυτά τα θέματα είναι θέματα για τα οποία κυρίως αρμόδια είναι τα κράτη-μέλη. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το πολύ κάτι συμπληρωματικό. Από την άλλη μεριά, όπως προτείνει και ο εισηγητής και ο κ. Κοσλόφσκι, πρέπει να προσπαθήσουμε τα μέσα που έχει η Ένωση στη διάθεσή της να είναι πιο αποτελεσματικά στην καταπολέμηση αυτή της ένδυας. Κύριε Κοσολίνο, θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Κοσλόφσκι. Όχι, συμμερίζομαι τα, τα περισσότερα από αυτά που είπε, θα προσπαθήσουμε να εργαστούμε και να παρουσιάσουμε μια κοινή πρόταση τη Επιτροπή Προπολογισμών. Πολύ καλά. Επ' αυτού θα ήταν έξοχο κάτι τέτοιο, λέει ο Πρόεδρο. Υπενθυμίζω το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για τι τροπολογίε 21 Ιουνίου. Προβλέψαμε την έγκριση του σχεδίου γνωμοδοτήσεω στη συνεδρίαση τη Επιτροπή Προπολογισμών στι 12 και 13 Ιουλίου, ούτω ώστε η Επιτροπή Απασχόληση να διαφωτιστεί από την γνωμοδότησή μα για την ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Απασχόλησης στις 8 Σεπτεμβρίου. Ιδού, λοιπόν, σας προτείνω τώρα να δώσουμε το λόγο στο Λάσλο Σούριαν όσον αφορά το σημείο 11, το σχέδιο γνωμοδότησής του όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι μια γνωμοδότηση που θα υποβάλουμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, η οποία εξέφρασε την επιθυμία να ετοιμάσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Αρκετά σημαντικό λοιπόν το θέμα. Ε, Λάσλο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικό ζήτημα πράγματι. Ε, συμφωνώ με αυτή την άποψη. Όμως Εάν θέλουμε να δούμε με κριτικό μάτι το θέμα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη προσέγγιση. Πρέπει να παραμείνουμε στο πλαίσιο της επιτροπής προϋπολογισμών. Άρα περιορίζεται και η γνωμοδότησή μας και η άποψη θα εκφράσουμε από το πλαίσιο της Επιτροπής μας. δεν είναι και τόσο εύκολο και αστείο να προτείνει στην Επιτροπή να αποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένη ημερομηνία, συγκεκριμένο υλικό. Δεν μπορούμε να προτείνουμε εμεί στην Επιτροπή την οικονομική πώ να κινηθεί. Εμεί πρέπει να κοιτάμε τα δικά μα και αυτοί τα δικά του. Στη σύντομη αυτή γνωμοδότηση λοιπόν επικεντρώνομαι επί πέντε παραγράφων. Και θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Χρονισμός. Το πρώτο κομμάτι του έτους πρέπει να επικεντρωθεί η διαδικασία. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλω να τονίσω. Αρχές του έτους. Μετά χρειάζεται συνεργασία συνεργασία ε, μεταξύ ε, εθνικών προϋπολογισμών και κοινοτικού. Τρίτον, θέλουμε να παραμείνουν διακοινοβουλευτικές ε, συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα ετησίως. Είναι και χειρονομία ευγενίας αν θέλετε, αλλά καμιά φορά είναι και σημαντικές και χρήσιμες αυτές οι συναντήσεις. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μας δίνει πράγματι ένα θέμα για τις διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την ε, πρακτική που ακολουθούμε. Στο σημείο 4 αναφερόμαστε στο κείμενο αυτό στην ε, πολιτική συνοχής. Άκουσα κάποιες επικρίσεις για αυτό. Γιατί αναφέρουμε μόνο, λέει, το, την πολιτική συνοχή στο έγγραφο. Αυτό μου είπαν. Είναι βασικό εργαλείο η πολιτική συνοχή για τη στρατηγική του 2020. Και γι' αυτό πρέπει να αναφέρεται. Και άλλα τμήματα του προπολογισμού δεν είναι τόσο σχετικά για, την, ε, για το σκόπο αυτό. Εάν λάβω υπολογίε θα προσπαθήσω να κάνω παραχωρήσεις για να έχω την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Όπως και την προηγούμενη φορά που αναφέρθηκα στις δυνατότητες που έχει αυτή η γνωμοδότηση, έτσι και τώρα λέω ότι πρέπει να σεβαστούμε κάποιες ευαισθησίες. Το βασικό είναι ότι το εξάμεινο αφορά περισσότερο Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το μήνυμα που βγαίνει από την Οικονομική Επιτροπή είναι ότι το Κοινοβούλιο αποτελεί ένα απόσταστο τμήμα τη διαδικασία. Και εμεί, σαν Επιτροπή Προπολογισμών, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Πρέπει να συμμετάσχουμε και εμεί στη διαδικασία. Τουλάχιστον αποκτώντα πληροφορίε. Και μετά μαζί με τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να δούμε τι ποσά χρησιμοποιούνται για τους στόχους του 2020 στον εθνικό προπολογισμό, στους εθνικούς προπολογισμού. πώς μπορούμε να βοηθήσουμε οι μεν τους δε όσον αφορά θέματα προπολογισμού. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν Πρόεδρε, αυτή είναι η πρόταση. Είμαι ανοιχτό για συζητήσεις με τους κοιόδης ηγητές και με άλλους που ενδιαφέρονται για το θέμα και αν θυμάμαι σωστά την περασμένη φορά σας έδωσα ένα χρονοδιάγραμμα ήταν στο Κόμπου News. Έχουμε περίπου μία εβδομάδα για την υποβολή τροπολογιών. Και για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το έργο μας. Ακούγονται φήμες στον τύπο κυρίως ότι υπάρχει κάποια ένταση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου. Αυτό δεν μας αφορά. Δεν με χαροποιεί αυτό. έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατανόησε τις επιθυμίες των κρατών μελών για αυτή τη διαδικασία, που την ξεκίνησαν τα κράτη-μέλη. Και αφορά εθελοντική συνεργασία στον τομέα της οικονομικής πολιτικής. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καμιά φορά συμπεριφέρεται σαν δάσκαλος, που διδάσκει τους μαθητές και τιμωρεί τα κράτη-μέλη τους μαθητές. Το είπε και ο Επίτροπο όσον αφορά το μέλλον. Το μέλλον τη διαδικασία είναι στα χέρια των κρατών μελών. Αυτά ξεκίνησαν τη διαδικασία, αυτά πρέπει να κάνουν τη δουλειά του. Να δούμε πόσο θέλουν την εναρμόνιση τη οικονομική πολιτική, των οικονομικών πολιτικών. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Τα θέματα του υπολογισμού είναι κάπω στο περιθώριο. Η θέση μα είναι αρκετά απλή. Δεν θα ανακατευτούμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Μπορούμε απλώς να λυπούμαστε να χαιρόμαστε για αυτά. Εγώ λυπούμαι λίγο, ελπίζω να με υποστηρίξουν και οι άλλες ομάδες. Πολύ καλά. Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά για την παρουσίασή σας και τη σαφέστατη παρουσίαση της θέσης σας. Νομίζω πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα Και είναι θεμητό η Επιτροπή Προπολογισμών να κάνει τις προτάσεις της. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα σε δύο ζητήματα, τα οποία ήδη συμπεριλαμβάνονται στο κείμενό σας, αλλά θα μπορούσαν να συμπληρωθούν ή να βελτιωθούν. Αν θέλετε, μπορούμε να συνεργαστούμε γι' αυτό και μαζί με τους άλλους σκιώδες και τους συντονιστές. Πρώτον, να προτείνουμε ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να αποτελεί στοιχείο της ε, διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Ο εισηγητή, η εισηγήτριά μας ε, για τον προϋπολογισμό του 2012, η κυρία Μπαλτσάνη, μας το πρότεινε και το δεχτήκαμε. Ήταν μια ιδέα για τον προϋπολογισμό του 2012 που είναι πάρα πολύ σημαντική ήδη από τώρα. γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένος και με πρωτοβουλία της Επιτροπής Προπολογισμών έχει εκφράσει την επιθυμία του η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου η διαδικασία δηλαδή καλύτερου συντονισμού των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών να μην περιορίζεται στην εξέταση μόνο στην καταπολέμηση των ελλημάτων και του χρέους αλλά να επεκταθεί και στο να επεκτείνεται και στο περιεχόμενο των εθνικών προπολογισμών προκειμένου να εξασφαλιστεί, να εξασφαλίζεται τακτικά κάθε χρόνο ότι οι εθνικοί προπολογισμοί λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της ε, Ευρώπης 2020. Όλοι τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν εξοικονομήσεις, να μειώσουν τις δαπάνες τους, να μειώσουν τα έλλειμματά τους. Αλλά ταυτόχρονα έχουν αναλάβει τη δέσμευση να πετύχουν τους στόχους της Ευρώπης 2020. Και όλοι θα πρέπει να συμμετάσχουν ε, στο μερίδιο που τη αναλογεί στη χρηματοδότηση τη Ευρώπη 2020. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Δημοσιονομική Πειθαρχία και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο όμω γινόταν λόγο μόνο για τα ελλείμματα. Στο τελευταίο Συμβούλιο Κορυφή όμω, Μαρτίου, Απρίλιο, δεν θυμάμαι πότε ήταν, εισήχθη και ο στόχος ο πρόσθετος στόχος στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας να αξιολογείται και η καλή υλοποίηση των στόχων της Ευρώπης 2020. Αν λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέχεται αυτή την καινούρια διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τότε ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμό σίγουρα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Γιατί? Γιατί τουλάχιστον το 50%, αν όχι το 60% του ευρωπαϊκού προπολογισμού αφιερώνεται στην Ευρώπη 2020. Και αυτό το ποσοστό ίσως θα αυξηθεί στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί η Επιτροπή Σούρε στην έκθεσή της καθιστά την Ευρώπη 2020 ε, βασική αναφορά, πυλώνα, σπονδυλική στήλη της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Συνεπώς, αν γίνει δεκτή αυτή η ιδέα, θα έχει και παιδαγωγική δράση, ε, διδακτική δηλαδή, θα είναι διδακτική και, στα για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ε, στα, μεταξύ των οκτώ ε, προϋπολογισμών που ε, εξετάζονται, μόνο ένας, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, είναι πάντοτε ισοσκελισμένος. Και ένα μεγάλο κομμάτι του ε, αφιερώνεται στην Ευρώπη του 2020. Συνεπώς, η όλη αυτή διαδικασία θα ε, μας βοηθήσει να δείξουμε στους υπουργούς οικονομικών και στους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων την ιδιαιτερότητα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Γιατί σήμερα ε, έχουν την εντύπωση ότι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι παρόμοιο με ε, τους εθνικούς Όχι, είναι ένας ιδιαίτερος προπολογισμό με πολύ μικρές ποσοστιά δαπάνες, πολύ μικρότερες από τους, ευρωπαϊκούς, από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και μια σειρά δράσεων στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 πολύ σημαντικών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώ, ο προπολογισμό αυτός θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και θέλουμε εμείς να είμαστε ο 28ος συμμετέχων. Ε, το άλλο που ανέφερε ο Λάσλο, η παρέμβαση των κοινοβουλίων στην όλη διαδικασία των Εθνικών Κοινοβουλίων και αν ε, συμπεριληφθεί και ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός και το, και το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια καινούργια ιδέα. Είμαστε οι πρώτοι που την υποστηρίζουμε και έχουμε λάβει την υποστήριξη και κάποιων Εθνικών Κοινοβουλίων επίσης. Ε, το θέμα αυτό ήταν κεντρικό στην συζήτηση ε, του περασμένου Απριλίου με, τους, ε, με τις Επιτροπές Προεπολογισμού των Εθνικών Κοινοβουλίων, με τις οποίες συναντηθήκαμε εδώ στις ε, Βρυξέλλες. Και θυμάστε ότι όλες, όλα τα κοινοβούλια ενδιαφέρθηκαν για αυτή την ιδέα, δηλαδή να μπορέσουν να συμμετάσχουν και στην διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμείνου. Δύο είναι οι τρόποι συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων, οι δύο δυνατότητες. Πρώτον, ε, μέσω μιας εσωτερικής εθνικής διαδικασίας το ε, κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο να προσπαθήσει να ζητήσει από την αντίστοιχη κυβέρνηση να συμμετάσχει στην διαδικασία προετοιμασίας της ε, χώρας για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σε ό,τι αφορά τον, ε, τον εθνικό προπολογισμό. Αυτό γίνεται ήδη στην πλειοψηφία των χωρών, είναι κάτι φυσιολογικό. Ο δεύτερος τρόπος συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων θα ήταν ο εξής, να πάρουν μέρος στις ίδιες τις συζητήσεις που γίνονται στις ευρωπαϊκές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο μιας διακοινοβουλευτικής συνάντησης. Αυτή η ιδέα ε, συγκέντρωση των ενδιαφέρον των Εθνικών Κοινοβουλίων τον Απρίλιο και πιστεύω ότι ε, είναι μια καλή ιδέα. Διότι αν δεν ε, λάβουν μέρος πλήρως όλα τα εθνικά κοινοβούλια από την πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αυτή η διαδικασία δεν θα λειτουργήσει. Αν δηλαδή η διαδικασία αυτή αφορά μόνο τους μοιημένους, τους συνήθεις υπόπτους, τους Υπουργούς Οικονομικών, την Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών, το ΚΟΡΕΠΕΡ και μια γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Η πολιτική νομιμοποίηση αυτής της διαδικασίας θα είναι πολύ ισχνή. Δεν θα γίνει δεκτή δηλαδή από τα κράτη μέλη, από τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, από τα μέσα και από την εθνική κοινή γνώμη. Οπότε οι ιδέες της Επιτροπής μας ε, είναι κρίσιμες. Ε, οι συνάδελφοι της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων από την άλλη μεριά ενδιαφέρονται πιο πολύ για το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει το Κοινοβούλιο ε, στην επιτήρηση, ε, στην εποπτεία των όσων συμβαίνουν στα κράτη-μέλη. Το λέω έτσι σχηματικά. Όμως η δική μας πρόσθετη προσθέμενη αξία ε, θα έπρεπε να είναι ότι πρέπει να καταδειχθεί πως το θέμα δεν είναι εμείς να ελέγχουμε πολιτικά το τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Όχι. Ο δικό μα ρόλο είναι να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν υπόψη στην εθνική του πολιτική πλήρω τους ευρωπαϊκού στόχου, του οποίου έχουν ήδη δεχτεί. Ο βασικό σημερινό στόχο, που είναι η, ο μηδενισμό των ε, δημοσιονομικών ελλημάτων, αλλά ταυτόχρονα πιο μακροπρόθεσμα ο στόχος μας είναι επίσης να χρηματοδοτήσουμε και τα μεγάλα project της ε, Ευρώπης 2020. Με αυτόν τον τρόπο ε, θα γίνουμε και πιο διδακτικοί σε ό,τι αφορά ε, την... και πιο πιστικοί σε ό,τι αφορά το το αίτημά μας ε, να διατηρηθεί ο προπολογισμό μας σε κάποιο συγκεκριμένο ύψος στα έτη 2014-2020. Διότι αν δοθεί προτεραιότητα μόνον στην δημοσιονομική πειθαρχία, ε, καταλαβαίνετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και εμείς και η Επιτροπή Σούρε ζητούμε να, να ε, ε, υπάρξουν εγγύησεις για μια μικρή αλλά σταθερή αύξηση του προπολογισμού, του ευρωπαϊκού προπολογισμού μετά το 2014, έτσι ώστε να βγούμε από την οικονομική κρίση και όταν βγούμε από την οικονομική κρίση να ε, έχουμε επαρκείς πόρους για να χρηματοδοτήσουμε τις επενδύσεις. Συνεπώς είναι, ε, η κίνηση αυτή θα είναι διδακτική, θα έχει ένα, έχει να παίξει ένα παιδαγωγικό ρόλο έναντι των ε, εθνικών κυβερνήσεων. Και έναντι βέβαια της ε, άποψης της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Ας βρούμε την πιο κατάλληλη διατύπωση αυτής της ιδέας. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, θα... Ε, α, μας μένει ένα τελευταίο θέμα ουσίας που θα πρέπει να εξετάσουμε σήμερα το απόγευμα. Ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση του κ. Αλφόνση για την πολύ ενδιαφέρουσα ε, το πολύ ενδιαφέρον θέμα τη Συμφωνίας Ευρωπαϊκή Ένωση με το Πράσινο Ακροτήριο σε θέματα αλίας και βέβαια έχουμε και τον Αντιπρόεδρο τη Σερβικής Κυβέρνησης καθώς επίσης και μια τελευταία ψηφοφορία για την έκθεση Ματέρα. Νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε τι εργασίε μας εδώ το πρωί και το απόγευμα η συνεδρία σήμερα θα είναι αρκετά light πρότεινα στον αντιπρόεδρο της ε, σερβικής κυβέρνησης να έρθει λίγο πιο νωρίς από το είχαμε προβλέψει αρχικά. Μπορεί να έρθει από τις 4 παρατέταρτο και μετά. Οπότε σας προτείνω να ξεκινήσουμε στις 3 και 4, 3 και 4 ξανά. Θα στείλουμε ένα mail σε όλα τα μέλη για να τα ενημερώσουμε για αυτή την καθυστερημένη έναρξη της συνεδρίασης. Ε, θα ξεκινήσουμε την έκθεση Αλφόνση. Μετά από τις 4 παρατέταρτο και μετά θα συναντούμε τον αντιπρόεδρο της σερβικής κυβέρνησης. Θα μας αφιερώσει μία ώρα περίπου και θα ψηφίσουμε την ε, έκθεση Ματέρα αμέσω μετά. Θα ήθελα να είναι παρόντες όσο να το περισσότερο συνάλφη για λόγους ευγένεια, προφανώς, και ε, προκειμένου να εξασφαλίσουμε απαρτία στην ψηφοφορία. Σίγουρα θα τελειώσουμε πριν τις 6.30. Ευχαριστώ πολύ. Διακόπτουμε.